Guten Morgen. Ähm, Bitte nehmen Sie Platz. Ich bin hier über die Fransen gefahren. Ja, wir, ich eröffne die Sitzung der Haushaltskontrolle leicht verspätet. Tut mir leid, aber es sind. Ξεκινάμε λίγο καθυστερημένα. Η ημερήσια διάταξη σας έχει κατατεθεί. Εξ όσων γνωρίζω ε, δεν υπάρχουν επιτιμίες για αλλαγέ. Πάμε στο σημείο υπαρτιμών 2 της ημερήσιας διάταξης να σας επισημάνω το γλωσσικό καθεστώς και εκτός αυτού θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε και δανέζικα και ρουμανικά. Η συζήτηση και η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου, ο συνήθως, και θα ήθελα να έχετε κατά νου ότι αν λάβει το λόγο θα ε, είναι και η κάμερα στραμμένη προς εσάς. Τα πρακτικά τα έχετε μπροστά σας. Εάν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ε, ε, δεν έχετε καταθέσει προσφυγή για τα πρακτικά, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 4 της ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ, για την υπόθεσή του από την τελευταία φορά που είχαμε αναβάλει. Παρακαλώ, κύριε Μαριά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι προσωπική υπόθεση, απλά βλέποντας τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την ε, <clears throat> πρόσληψη ε, τοπικού ε, προσωπικού, local assistance, θα ήθελα να κάνω κάποια πρόταση, να τη λάβουμε υπόψη, ούτως ώστε να έχουμε ίσως μια αλλαγή της διαδικασίας. η διαδικασία για την πρόσληψη ΑΠΑ είναι για μένα η καλύτερη, δηλαδή πρώτα υποβάλλεται η αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται τα έγγραφα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εν συνεχεία όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογράφεται η σύμβαση. Επομένως υπάρχει μια σαφήνεια στο πώς λειτουργεί η διαδικασία. Για να προσληφθεί ένας ε, local assistant θα πρέπει, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, να υπογράψει μια σύμβαση με τον ε, Ευρωβουλευτή. Και φυσικά να τηρηθούν και οι διαδικασίες που έχουν σχέση με την εργατική νομοθεσία. Δηλαδή να ανακοινωθεί η πρόσληψη αυτή στις ε, τοπικές αρχές. Εν συνεχεία η διαδικασία ακολουθείται ως εξής. Γίνεται, φέρνουμε ε, τα έγγραφα στην ε, DG FINS προς έγκριση. Συνήθως εγκρίνονται. Εάν όμως δεν εγκριθεί η διαδικασία αυτή, τότε συμβαίνει το εξής παράδοξο. Να έχει αναλυφθεί μεν μια υποχρέωση του Ευρωβουλευτή απέναντι στον local assistant και ως εκ τούτου ο Ευρωβουλευτής να είναι υποχρεωμένος να του καταβάλει τους μισθούς και τις ασφαλιστικές φορές και από την άλλη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην εγκρίνει την πρόσληψη αυτή. Και επειδή διαρκεί αυτό τουλάχιστον 20 μέρες με 25, αντιλαμβάνεστε ότι οι εξουσίες μεν είναι στην DG να εγκρίνει το συμβόλαιο, αλλά οι υποχρεώσεις είναι μονομερές, μόνο στον Ευρωβουλευτή. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι χρειάζεται μια αλλαγή της διαδικασίας. Εγώ θα προτιμούσα να κάνουμε αυτό που συμβαίνει με τους ΣΑΠΑ, δηλαδή να, γίνεται, να φέρνουμε τα έγγραφα, να εγκρίνονται και από τη στιγμή που εγκρίνονται από την DGFINS τότε να υπογράφεται και η σύμβαση. Διότι δεν μπορεί να εγκριθεί η πρόσληψη local assistant από την DGFINS εάν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση. Δεύτερο, θα ήθελα να δούμε και το θέμα του paying agent Δηλαδή επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ή άλλως έχει γραφεία σε όλε τι χώρε, θεωρώ ότι η αλλω εχει γραφεια σε ολε τι χωρε θεωρω οτι η καλυτερη διαδικασια θα ήταν να πληρώνονται απευθεία και οι local assistants από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι εύκολο αυτό όσον αφορά του μισθού, διότι μπορούν να δώσουμε ένα λογαριασμό, η μισθή, το ύψο του μισθού είναι συγκεκριμένο και να πληρώνονται. Το πρόβλημα είναι ίσω με τι ασφαλιστικέ εισφορές και του φόρου που πρέπει να πληρώνεται σε κάθε κράτο. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να το δει και να μας βοηθήσει I'm going to finish, Madam President. Θα μπορούσε να μας βοηθήσουν τα τοπικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί και εκεί έχουν staff και πληρώνουν ασφαλιστικές φορές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να το δούμε σοβαρά, διότι ο paying agent αναλαμβάνει να πληρώσει, αλλά καμιά φορά είναι δυνατόν να μην πληρώσει ο paying agent ή να πτωχεύσει ή να του κατάσχουν λογαριασμούς. Οπότε τότε πάλι υπεύθυνο είναι ο ευρωβουλευτής να πληρώσει τους μισθούς, ενώ δεν έχει καμία ευθύνη. Θέλω λοιπόν στο πλαίσιο της διαφάνειας να συνδυαστεί αυτό και με την υπευθυνότητα. Να έχουμε ευθύνη όταν έχουμε εξουσία. Όταν δεν έχουμε εξουσία δεν μπορούμε να έχουμε ευθύνη. Σας το θέτω υπόψη αυτό. Χτες ψηφίσαμε μερικές αλλαγές για τον τρόπο λειτουργίας των προνομίων και των εξουσιών του Ευρωβουλευτή και επομένως αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε με έναν προβληματισμό ε, για το πώς θα μπορούσε ενδεχόμενα να αλλάξει η διαδικασία πρόσληψης των τοπικών βοηθών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ähm, Αυτές οι διαδικασίες, ξέρετε, έχουν προκύψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό γιατί το 2009 υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ λέω το εξής, αυτό το όλο θέμα βεβαίως και θα το συζητήσουμε με τη διοίκηση του Κοινοβουλίου αλλά θέλω να επισημάνω ότι ε, τα γραφεία στις ε, πρωτεύουσε έχουν ε, ειδικού επικοινωνίες και όχι ειδικού για θέματα οικονομικά. Αυτό που προτείνετε εσείς ξέρετε τι θα σήμαινε. Θα σήμαινε τεράστια αύξηση του προϋπολογισμού και του προσωπικού και αυτό εγώ δεν το βρίσκω απαραίτητα σωστό. Δηλαδή αυτά δεν μπορεί κανείς να τα αποφασίσει εν μια νυχτή. καλύτερα να αφήσουμε λίγο χρόνο και πιστεύω ότι είναι καλή καλύτερα να δώσουν δυνατότητα να συζητηθεί το θέμα με τη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Εντάξει, το λαμβάνουμε υπόψη μα, αλλά προ το παρόν δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε στο θέμα. Και παρακαλώ κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, εγώ ε, το έθεσα ω προβληματισμό. Δεν είπα να πάρουμε απόφαση σήμερα. Είναι κάτι που μα απασχολεί, αλλά τουλάχιστον να τεθεί, να το συζητήσουμε με ηρεμία με τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να υπάρξει μια λύση. Δηλαδή, θα έχουμε ευθύνη όταν έχουμε και εξουσία. Όταν δεν έχουμε εξουσία δεν μπορούμε να έχουμε ευθύνε. Α δούμε έναν τρόπο, ευχαριστώ πολύ που το λάβατε υπόψη και να δούμε πώ θα το συζητήσουμε με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ευχαρίστω θα το κάνω κύριε Μαριά. Πάμε τώρα στο σημείο υπερθμών 4 τη ημερήσια διάταξη. Ε, που είναι η κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού τα καλωσορίζω θερμά και πρέπει να ε, γίνει κάποια παρουσίαση. Έχουμε τον συνάδελφο από την Επιτροπή Προϋπολογισμού και εγώ από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τους τελευταίους τριμερείς διαλόγους όπου συμμετείχαν κάποια θαραλέα ε, μέλη εξημών. Να σας πω λοιπόν ότι στις 16 ε, και στις 25 Νοεμβρίου, λέει η Πρόεδρος, ε, είχαμε τριλόγους. Ε, θέλω να σας επισημάνω ότι υπάρχουν 270 άρθρα με πάρα πολλές αλλαγές. Έτσι λοιπόν 16 Οκτωβρίου διερθώνει τώρα η Πρόεδρος, 16 Οκτωβρίου Πλέον έχουμε νέα διατύπωση από την Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, για τα άρθρα 3 μέχρι 81 και έχουμε φτάσει μέχρι το άρθρο 114 και τώρα πλέον συμφωνήσαμε ότι το 59.1 άρθρο 59 για τη σύγκρουση συμφερόντων όπως και το 61AC παράγραφος 2 62 δεύτερο εντάφιο ΧΑ επ' αυτού καταλήξαμε σε συμφωνία και κατά τα άλλα ε, συμφωνήσαμε και για τα άρθρα 68, 69, 2, 72 και 73. Δηλαδή και για το θέμα του sponsoring, για τον ορισμό των ε, επιδομάτων και για τα ε, Regie d'Avance στα γαλλικά, που ψάχνω να βρω το γερμανικό ρόλο, δεν τον βρίσκω, και για την Regie d'Avance μπορέσαμε να βρούμε έναν, ε, μια συμφωνία για το άρθρο 58-56. Έχουμε το 69-6 ε, για τον έλεγχο των ε, ε, γραφείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης τα άρθρα 31-2, 32-3, 33-1, 73-2 σχετικά με το τι είναι performance όπως λέει αγγλικά, ποιοι είναι οι δείκτες απόδοσης και πώς μπορούμε να εντάξουμε αυτούς τους δείκτες ε, στον προϋπολογισμό. Ε, επ' αυτών δεν έχουμε ακόμα συμφωνήσει και δεν έχουμε συμφωνήσει και για τον ορισμό στο άρθρο 2 του 27. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί αφορά χρηματοδοτικά εργαλεία και αφορά επίσης ε, και τα revolving funds, τον σχετικό ορισμό. Εξάλλου δεν έχουμε λύση και αυτό ε, που ορίζει η Κομισιόν ως ε, μαξιλάρι ευελιξίας. Ε, κάτι άλλο. Δεν έχουμε λύση και το θέμα της ανάθεσης ε, αρμοδιοτήτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλους θεσμούς. Ε, το θέμα κυρίως ε, πώς ενημερωνόμεθα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κατά τα, επόμενα έτη θα πρέπει να θεωρούμε ότι θα υπάρχουν μεγάλες αντιπροσωπείες. Και δεν έχουμε συμφωνήσει και για την διαφάνεια των αποδεκτών επιδοτήσεων για, το, για τους συντελεστές, τους πολλαπλασιαστές κυρίως όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις. Εχθές λοιπόν από το άρθρο 115 φτάσαμε στο άρθρο 170 περίπου. Ε, δεν συμφωνήσαμε σε όλα, αλλά νομίζω εχθές μπορούσαμε να κλείσουμε τα 115, 17, 18, 21, 22. εκεί ε, το Κοινοβούλιο συμφώνησε και ε, θέλω να σας πω ότι τελικά ενδώσαμε Cross Alliance έχουμε στο άρθρο 23, στο 24, στο 28 μέχρι 131 μέχρι και το 171 για όλα αυτά συμφωνήσαμε Δηλαδή για τα υπόλοιπα υπάρχουν νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε θέματα τα οποία είναι σημαντικά της Επιτροπής Προπολογισμού και της Ελέγχου Προπολογισμού, όπως η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου ή τα θέματα των εικονικών εταιριών, επ' αυτών εξακολουθούμε να έχουμε κάποια ανοιχτά σημεία. Ανοιχτό παραμένει και το θέμα του εφάπαξ ποσού ε, και στον ορισμό και στη διαπίστωση. Όσον αφορά τις εφάπαξ ε, δαπάνες, ε, νομίζω ότι εκεί χρειαζόμαστε ακόμα κάποιες διευκρινήσεις. Όπως σας είπα, δεν τα ρυθμίσαμε όλα αυτά γιατί δεν είχαμε αρκετό χρόνο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 in terms of timescale, I think if we were optimistic, we would say that we would probably finish by the end of December. Thank you. Ja, besten Dank. Die Frau Kollegin Ayala, bitte. Ευχαριστώ, κυρία Ayala. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για τα όσα μας είπατε και για την ενημέρωση που μας κάνατε. Θα ήθελα να ζητήσω κάποια διευκρίνηση όσον αφορά το ε, θέμα ότι μπορεί να είμαστε όμοιροι άλλων ε, κανόνων όπως ας πούμε είναι το Connecting Europe, αυτή η διευκόλυνση. Ε, βεβαίως ε, όσον αφορά τα συγκεκριμένα στοιχεία είχα καταλάβει την τελευταία φορά που μας ενημερώσατε κυρία Πρόεδρε ότι υπήρχε δυνατότητα τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι κανονισμοί να ε, δημιουργηθούν νωρίτερα και επομένως ε, να πιέσουν ε, και εμάς στη δική μας περίπτωση. Τώρα λίγο ησύχασα γιατί καταλαβαίνω ότι δεν θα μας πιέσουν όλοι οι σύντροφοι και οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι σας για το θέμα αυτό. γιατί εγώ αυτό που θα ήθελα θα είναι να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε έναν ε, κανονικό καλό ρυθμό ε, χωρίς ε, να έχουμε εκνευρισμό γιατί μας πιέζουν οι συνάδελφοι. Δηλαδή να αφήσουμε τους άλλους να ψηφίσουν και να προχωρήσουν και εμείς να προχωρήσουμε με τον δικό μας ρυθμό ξεκαθαρίζοντας σε βάθος όλα τα στοιχεία. το πρόβλημα είναι... ότι ε, στους ε, άλλους ε, κανονισμούς. Ε, έχουμε ένα άρθρο στο τέλος και βάσει αυτών λειτουργούμε. Περιμένουμε λοιπόν το Συμβούλιο, πώς θα αποφασίσει το Συμβούλιο δεν ισχύει το ότι όλα έχουν ξεκαθαριστεί στο Συμβούλιο. Θα μιλήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και θα δούμε και πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα νομικά. Αλλά το θέμα είναι ότι ε, τον ε, Νοέμβρη πίστευε η Κομισιόν ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα και αν ε, κρατήσουμε αυτή την ταχύτητα νομίζω θα τα καταφέρουμε. Τελικά βέβαια ενδεχομένως θα κατορθώσουμε όλα αυτά τα θέματα να τα επιλύσουμε μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποια θέματα αρχής επί των οποίων δεν έχουμε συμφωνήσει. Ως εκ τούτου την εβδομάδα του Νοεμβρίου. 7 και 8 Νοεμβρίου θα έχουμε ε, δύο ε, τριμερείς διαλόγους ε, που θα διαρκέσουν πολύ και νομίζω εκεί θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Και βεβαίως ε, αυτό που θα χρειαστεί είναι να καθορίσουμε τις πολιτικές γραμμές. Πάντως, χωρίς την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και χωρίς να υπάρξει σχετική ψηφοφορία, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει μία αίτηση και την επόμενη εβδομάδα ή αν θέλετε την αποκαλούμενη πράσινη εβδομάδα θα μπορέσουμε να καταθέσουμε αυτό το αίτημα. Πιστεύω λοιπόν ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει. Δεν είναι δικό μας, δεν είναι δική μας η ότι χρειαστήκαμε τόσο χρόνο. Ε, ξεκινήσαμε καθυστερημένα γιατί το Συμβούλιο χρειάστηκε περισσότερο χρόνο. Έχουμε 127 ε, τροπολογίες και ως ε, εκ τούτου ε, θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ε, διαπραγματευτούμε, να αντιπαρτευτούμε με τους υπόλοιπους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν τελικά εκείνη επιθυμεί να προχωρήσουμε, θα πρέπει και αυτό να αποφασιστεί ομόφωνα στο Συμβούλιο. Ως εκ τούτου ε, δεν θα ήθελα να στριμώξω κάθε έναν από τους ενδιαφερόμενους και να τους αναγκάσω να προχωρήσουν. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε ακόμα τουλάχιστον όσον αφορά αυτά τα θέματα μέχρι τον Ιανουάριο να τα διασφαλίσουμε και ε, το θέμα του προπολογισμού σίγουρα δεν θα μπορέσει να τεθεί τον Ιανουάριο γιατί χρειαζόμαστε ακόμα πάρα πολύ χρόνο με τους ε, νομομαθείς. Υπάρχουν ακόμα ελπίδες αλλά από την άλλη θεωρώ ότι και μπορεί να αρχίσει να ισχύει και το άρθρο 167. Θα τηλεφωνήσουμε πάρα πολύ, θα μιλήσουμε πάρα πολύ, αλλά υπάρχει ελπίδα ε, στις επόμενες, στους επόμενους δύο τρι, τριμερείς διαλόγους να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά. Αυτά είχα να σας πω και έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του σημείου της μέσης διάταξης. Αν δεν έχετε άλλες ε, παρατηρήσεις, θα έλεγα να περάσουμε στο σημείο υπαριθμών 5 της σημερινής διάταξης. Ε, είναι μια έκθεση πρωτοβουλία ε, του συναντέλφου Βόνο, ο οποίος ε, θα έχει και το λόγο για να μας παρουσιάσει ακριβώς αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Έχουμε πολλές εκθέσεις για το ίδιο θέμα. Έχουμε μια έκθεση ECA Ε, και αυτή είναι η δεύτερη γνωμοδότηση, αυτή είναι η δεύτερη έκθεση. Είχαμε και άλλη μία ε, όσον αφορά την ε, πρωτοβουλία για τους νέους καθώς επίσης και το Youth Guarantee Scheme. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Αυτή η employment ε, η initiative έχει ξεκινήσει με πολύ αργό ε, ρυθμό Νομίζω ότι όλοι θεωρήσαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν είχαν την ε, δυνατότητα ή τις υποδομές ε, εξ αρχής ε, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και να υλοποιήσουν σωστά το πρόγραμμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως, παρότι ξεκίνησε αργά, έγιναν κάποιες βελτιώσεις και ευελπιστούμε ότι, μάλλον βλέπουμε ότι είναι μάλλον αποτελεσματικά. Ας πούμε, βλέπουμε ότι ε, ο μέσος όρος της ε, ενεργή ανεργίας κατέβηκε από το 23 στο 16, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι πάρα πολύ καλό ε, και επομένως φρονούμε πως έχει βοηθήσει σε πολλά κράτη-μέλη. Ωραία, πολλά καλά νέα, αλλά βεβαίως πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν ο, θέλουμε να μην σταματήσει η χρηματοδότηση το 2020 αλλά να συνεχίσει και να ε, ενταχθεί και στο επόμενο ε, πολιετές ε, πλαίσιο, στο επόμενο MFF και βεβαίως όσο περισσότερα στοιχεία έχουμε τόσο πιο καλά μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Νομίζω ότι με την έγκρισή σας ε, κυρία Πρόεδρε νομίζω ότι μπορώ να συμπεράνω γενικά ότι ήταν ένα καλό πρόγραμμα και ότι επομένως ε, θα πρέπει να ε, επεκταθεί όχι μόνο μέχρι το 2020 αλλά και μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών είναι η 10η Νοεμβρίου και στις 27 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ως εκ τούτου τέλειωσε και αυτό το θέμα της σημερινής διάταξης. Ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω τώρα να ε, φέρετε, να βρείτε τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Γιατί τώρα πάμε στο σημείο υπερθμών 6 της σημερινής διάταξης που είναι η ψηφοφορία για, τα αιτήματα σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Έχουν κατατεθεί αρκετές ε, τροπολογίες Και αυτό μας εξέπληξε, διότι δεν υπήρχε και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να κατατεθούν τροπολογίες. Να σας πω ότι ρώτησα και εγώ την διοίκηση κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ε, δύο τροπολογίες ε, κατατέθηκαν από τη διοίκηση, τη υιοθέτησα και κατά τα άλλα όσον αφορά τις ε, τροπολογίες ε, για το, ε, για το ελεγκτικό συνέδριο και την ΕΠΟ προσπαθήσαμε στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα να είμαστε δημιουργικοί, θελήσαμε να προβάλλουμε αιτήματα και αυτά που εγώ κατέθεσα ως ε, εισηγήτρια ε, πραγματικά ήταν ε, αποδεκτά. Δεν ξέρω, μπορούμε τώρα, πιστεύετε μπορούμε να ψηφίσουμε, πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν και θα ήθελα να παρακαλέσω καταρχήν να δούμε πόσα μέλη έχουμε. Που πατήστε ένα κουμπί, ποιον να είναι, για να δούμε αν μπορεί να ξεκινήσει η ψηφοφορία, να δούμε δηλαδή πόσες κάρτες έχουμε. 20.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 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και νομίζω ε, υπάρχει και η επιθυμία να ψηφίσουμε unblock συλλήβδην όλες τις ε, επόμενες ε, τροπολογίες μέχρι το 45, το, την τροπολογία 45. Α, όχι.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 Η 56 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 58 υπέρ κατά αποχές ε, έλεγχος ηλεκτρονική επαλήθευση για την 58 παρακαλώ. εγκρίνεται, η 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 11 υπέρ κατά απορρίπτεται, η 12 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επανήλθευση για την 12 παρακαλώ. Ολοκληρώθηκε η επαλήτευση, εγκρίνεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 Καταπίπτει η 15 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται η 16 η... μισό λεπτό. 15 την ψηφίσαμε, 16 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται η 17 είναι γλωσσική τροπολογία, η 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ως εκ τούτου ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Μήπως υπάρχει κάποιος στην αίθουσα που δεν έχει κάρτα. Όχι, από ό,τι βλέπω. Ως εκ τούτου έκλεισε και αυτό το θέμα τη ημερήσια διάταξης. Και περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξης, που είναι η ανανέωση, ε, με η ακρόαση των μελών του Ελεκτικού Συνεδρίου σχετικά με την παράταση της θητείας τους. Και θέλω να σε επισημάνω ότι εχθές σα έστειλα μία επιστολή. Μία επιστολή όπου ε, αναφέρεται ότι θα συζητήσουμε και γι' αυτό που την τελευταία φορά, δηλαδή την αναβολή της ε, ψηφοφορίας ε, στην Ολομέλεια. Και στο τέλος θέλω να ψηφίσουμε για να καταλήξουμε στο κατά πόσον ε, η ψηφοφορία θα γίνει τον Ιανουάριο ή όχι. Νομίζω σας έχει ε, τεθεί, σας έχει υποβληθεί η επιστολή. Όλα αυτά θα τα ψηφίσουμε μετά την ακρόαση. Φαντάζομαι συμφωνείτε με όλα αυτά. Θα προχωρήσουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και ξεκινάμε με την ακρόαση του Ισπανού, ε, του κυρίου... Μισό Τον είχα δει λίγο πριν από λίγο τον Ισπανό υποψήφιο. Δεν τον βλέπω όμως στην αίθουσα. Πρόεδρος, νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλημέρα σας. Εδώ και έξι χρόνια περίπου, πριν από έξι χρόνια, Εμφανίστηκα για πρώτη φορά ενώπιον της Επιτροπής σας ως το, ο, υποψήφιος για το ελεγκτικό συνέδριο. Είχα τότε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την επαγγελματική μου στρα, σταδιοδρομία και να εκφράσω πόσο δεσμευμένος νιώθω για να συμβάλλω στο μέλλον του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχω την τιμή σήμερα να σας ζητώ να ανανεώσετε τη θητεία μου. Έχετε το ενημερωμένο βιογραφικό μου σημείωμα όπου φαίνονται τα 30 και πλέον έτη που έχω υπηρετήσει ε, το δημόσιο συμφέρον και ε, περιλαμβάνει το βιογραφικό μου σημείωμα και μία σύνοψη της δουλειάς μου στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο τέταρτο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου που ασχολείται με τον έλεγχο των ε, θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση των αγορών, τον ανταγωνισμό στην οικονομία, την καινοτομία, τις υπηρεσίες και τους διάφορους οργανισμούς και φορείς της Ένωσης, καθώς και ό,τι έχει να κάνει με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Είχα την ευκαιρία να ε, τεθώ επικεφαλής ε, ελέγχων οικονομικών ποινικού χαρακτήρα ήμουν υπεύθυνο για τη σύνταξη διαφόρων εκθέσεων μεταξύ άλλων για τα, για τα ευρωπαϊκά σχολεία και για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω κάνει και πέντε ελέγχους για την απόδοση και αυτές οι εκθέσεις έχουν οδηγήσει στη βελτίωση του, της διαχείρισης και του ελέγχου του προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα τη τιμή να εμφανιστώ ενώπιον σας αλλά και ενώπιον άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου πάνω από 20 ε, φορές, ε, πάνω από 20 διαφορετικές περιπτώσεις και πιστεύω πραγματικά ότι συνέβαλα έτσι ώστε η δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου να καταστεί πολύ πιο εμφανής, πολύ πιο ορατή ακόμα και στη δική μου χώρα. Με τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται το ελεγκτικό συνέδριο έχει εξελίξει και την μεθοδολογία του και τα προϊόν των εργασιών του. Κάτι που χαρακτηρίζει ε, το ελεγκτικό συνέδριο είναι το γεγονός ότι δουλεύουμε ομαδικά σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης. Αν πρέπει ένα, σε ένα θέμα να σταθώ που με κάνει περισσότερο από όλα υπερήφανο είναι η δουλειά που έχει γίνει και που έχουμε κάνει για τον έλεγχο της διαχείρισης από πλευράς της Ένωσης της οικονομικής ε, κρίσης και χρηματοπιστωτικής. Έχουμε πάνω από 20 τέτοιου είδου ελέγχους που διενεργούμε και αυτό ήταν βασικό προηγούμενο για τη νέα διάρθρωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Σήμερα οι πόροι στο ελεγκτικό συνεδρίο κατανέμονται με ευέλικτο τρόπο ανάλογα με το πόσο σημαντικό είναι το εκάστοτε καθήκον που πρέπει να ε, διενεργηθεί. Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των ελέγχων απόδοσής μας και να είναι αυτή η έλεγχη πιο σχετική, καθώς και τα συμπεράσματα που, στα οποία καταλήγουμε, έτσι ώστε οι συστάσεις μας να έχουν πραγματικά θετικό αντίκτυπο. Είναι επίσης σημαντικό να εργαστούμε για να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με όλα τα θεσμικά όργανα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που τυχόν ενδιαφέρονται για την εργασία μας. Οι προκλήσει τι οποίε αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διακυβέρνηση, οικονομική ανάπτυξη, περιβάλλοντο, κλιματική αλλαγή, μεταναστευτικών ροών, δημογραφικών εξελίξεων ή και ασφάλεια, αποτελούν ε, και μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τον έλεγχο των οικονομικών του κράτους, των κρατών, του δημοσίου και το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένο για όλα αυτά. Θέλω να επαναλάβω ε, πόσο υπέρ είμαι του ελέγχου του δημοσίου συμφέροντος με ποιότητα, με ανεξαρτησία, με πίστη στο σύστημα της απόδοσης λογαριασμών, γιατί αυτό είναι αυτό που καλλιεργεί και ενθαρρύνει την πίστη και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στα ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ θερμά. Στη διάθεσή σας παραμένω για ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ότι πραγματικά τηρήσατε απόλυτα το χρόνο, μιλήσατε μόνο για πέντε λεπτά. Επόμενος... Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αξιότιμα μέλη του, αξιότιμο μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Έχω μια ερώτηση, ίσως είναι κάπως ασυνήθιστη. Θέλω όμως να σας ρωτήσω για την Ισπανική κυβέρνηση. Την περασμένη φορά μιλούσαμε για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων από το 86 η Ισπανία πάντα στέλνει άνδρα Πώς το εξηγείτε αυτό. Και δεύτερον, γνωρίζω πολύ καλά τις συνθήκες. Πιστεύετε όμως ότι 28 ελεγκτές χρειάζονται ή μπορεί να γίνει η δουλειά και με 14. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τάραντ για αυτές τις ερωτήσεις οι οποίες αποτελούν πραγματική πρόκληση. Θα έλεγα λοιπόν καταρχάς ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να εκπροσωπήσω και να μιλήσω επισήμως εξ ονόματος της ισπανικής κυβέρνησης, ούτε της παρούσας ούτε των προηγουμένων. Πόσο μάλλον να εξηγήσω τα πεπραγμένα της τότε ισπανική ε, κυβέρνησης πριν από 20 χρόνια. Εγώ είμαι εδώ γιατί έχω τη δική μου επαγγελματική στρατιοδρομία και διαδρομή. Όμως, σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι η εκπροσώπηση των φίλων στην Ισπανική κυβέρνηση, στο Ισπανικό Κοινοβούλιο, στην Ισπανική δημόσια ζωή, σίγουρα ε, είναι σε επίπεδα πολύ ικανοποιητικά. Θα έλεγα ότι και τα δύο φύλλα εκπροσωπούνται επαρκώ. Έχουμε ειδικέ διατάξεις στην εκλογική νομοθεσία, στον εκλογικό μας νόμο, για να έχουμε οπωσδήποτε μία εκπροσώπηση 40 και 60 για τις ε, βουλευτικές εκλογές. Νομίζω ότι η χώρα μου ενδιαφέρεται ιδιαίτερως για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και ότι έχει πετύχει ήδη πολλά σε αυτό το τομέα. Αλλά αυτή είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Δεν μπορώ να επισήμω να εκφράσω τη θέση της ισπανικής κυβέρνησης. Εγώ χαίρομαι που με διάλεξαν, που είμαι εδώ, που μπορώ να είμαι υποψήφιο για άλλη μια φορά, γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερο το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου και γιατί πιστεύω ακρατάντως ότι όλη αυτή η εμπειρία που έχω αποκομίσει, που έχω συλλέξει, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και βοηθητική. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο θέμα στο, το οποίο θέσατε έχει να κάνει με τη συνθήκη. Και όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν βάσει της συνθήκης. Και η συνθήκη προβλέπει, όπως γνωρίζετε και εσείς καλά, ότι θα έχουμε ανθρώπους από κάθε χώρα. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι πολιτικά θεσμικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τις δικές της ρυθμίσεις. Σε κάθε περίπτωση στο δικαστήριο και στο ελεγκτικό συνέδριο θα έλεγα ότι είμαστε πλήρως ισότιμοι εμείς οι 28 πλήρως ανεξάρτητη και ατομικά και συλλογικά. Όλοι μας, ανεξαρτήτως από τη χώρα από την οποία προερχόμαστε, συμβάλλουμε στη δουλειά του ε, ελεγκτικού συνεδρίου και νομίζω ότι αυτό λειτουργεί και δουλεύει καλά. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, ε, λειτουργεί ανατμήματα, έχει διαφορετικά τμήματα, έχουμε ρυθμίσεις ευελιξίας Τώρα, αν ο νομοθέτη και η συνθήκη αλλάξει τις ρυθμίσεις, τότε το ελεγκτικό συνέδριο θα λειτουργήσει και αυτό διαφορετικά. Και θα πρέπει αναλόγως να προσαρμόσουμε την ε, εργασία μας. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις από τον κύριο Τάραντ. Όχι, πήρα τις απαντήσεις μου. Ευχαριστώ. Στον κατάλογο των ομιλητών, ο κύριος Σαβάμα έχει ζητήσει τον λόγο. Ευχαριστώ. Το ΕΛΚ έχει δύο ερωτήσεις και θα ήθελα να τις μοιραστούμε μεταξύ των δύο μελών, εμού και της ε, ε, συναδέλφου. Λοιπόν, αν έπρεπε να αποφασίσετε εσείς ο ίδιος ποιοι θα ήταν οι τομεί στους οποίους θα έπρεπε το ελεκτικό συνέδριο να επικεντρώσει τις προσπάθειές του τα επόμενα 5-6 χρόνια. Ποιους θα διαλέγατε δύο τομείς μόνο επιγραμματικά. Ποιοι νομίζετε ότι είναι πιο σημαντικοί. Στη δουλειά του ελεκτικού συνεδρίου και ο Τόμας θα κάνει την επόμενη ερώτηση. Δική μου ερώτηση είναι η εξής. Πώς θα βελτιώσετε τη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου και προσωπικώς εσείς πώς ε, τον θα συνδέσετε τους ελέγχους με τις επιδόσεις και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και των επιδόσεων στην ετήσια έκθεση. Απάντηση. Κοιτάξτε, το ελεγκτικό συνέδριο έχει ήδη καθορίσει τις προτεραιότητες στην ε, στρατηγική που έχουμε καθορίσει για τα επόμενα χρόνια για το ελεγκτικό συνέδριο για το 2018 μέχρι και το 2020 για την τριετία αυτή έχουμε ε, θέσει ως προϋπόθεση να βελτιώσουμε την ετήσια έκθεση και να ενισχύσουμε ε, την ε, μέρημνά μας και το μέλημά μας για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Τώρα δύο τομείς πολιτικής που έχουν ενδιαφέρον και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση γιατί εμείς καθορίσαμε έξι στην στρατηγική μας. Εάν το νέο σύστημα ιεράρχησης και ορισμών των ε, καθηκόντων λειτουργεί. Τελικά πιστεύω ότι θα ευθυγραμμιστούμε πλήρως ε, στις επιδιώξεις μας με τις επιδιώξεις της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές και θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Έχουμε τα ενημερωτικά σημειώματα του Συμβουλίου της Επιτροπής για τις νέες προτεραιότητες, για τους νέους οικονομικούς κανονισμούς και θα ενταχθούν και νέες πολιτικές. Δύο τομείς όμως που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερως είναι οι εξής. Πρώτον, πρέπει να δουλέψουμε για να διασφαλίσουμε ότι η αρχή της ενότητας και της ακαιρεότητας του προϋπολογισμού προστατεύεται και κατοχυρώνεται, άρα δεν υπάρχουν κενά στη λογοδοσία ότι δηλαδή όλες οι οργανωτικές ρυθμίσεις και συμφωνίες καλύπτονται από κάποιον ανεξάρτητο έλεγχο όπως είναι αυτός του ελεγκτικού συνεδρίου και είναι πρόκληση αυτό μεγάλη γιατί επανειλημμένως έχουμε αναφέρει ότι υπάρχουν κενά στους ελέγχους στην αρμοδιότητα. Έχουμε νέες διακυβερνητικές συμφωνίες και χρειάζεται ένα σωστό πλαίσιο λογοδοσίας ε, για να είναι σωστή η η ευρωπαϊκή διαδικασία αλλά και για να βρίσκει δικαίωση η κοινή γνώμη. Και αυτό καταρχάς και δεύτερος τομέας είναι η αποδοτικότητα, οι επιδόσεις. Πώς θα καταλήξουμε σε συστάσεις που να βοηθούν πραγματικά. Και από εκεί και πέρα, το μέλλον της ετήσιας έκθεσης, ε, απαντώ στο δεύτερο ομιλητή. Δεν ξέρω αν έχω υπάρξει πολύ συγκεκριμένος, αλλά ε, διακόπτει ο βουλευτής. Ο Τόμας ε, έθεσε συγκεκριμένο ερώτημα για τον έλεγχο με βάση τις επιδόσεις και την απόδοση. Είναι ένας από τους δύο βασικούς τομείς για εσάς είπατε. Άρα μπορείτε να μας προσδιορίσετε πολύ συγκεκριμένα τι θα κάνετε για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ. Πρώτον, για το μέλλον της ετήσιας έκθεσης. Αυτό είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους. Ήδη κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σε αυτό το τομέα. Έχουμε τις 35 συστάσεις στην τελευταία ετήσια έκθεση και νομίζω ότι πλέον είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τη δουλειά με βάση την προηγούμενη δουλειά τους ε, πόρους που έχουμε εξασφαλίσει. Δουλεύουμε σε τεχνικό επίπεδο με την Επιτροπή και τους εταίρους μας. Και νομίζω ότι η ετήσια έκθεση θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν εναλλακτικέ. Για παράδειγμα, να βασιστούμε περισσότερο στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, την οποία βεβαίως θα έχουμε ελέγξει και εμείς ε, πολύ προσεκτικά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα. Αυτό είναι πρόκληση, αλλά είναι και δέσμευση του ελεγκτικού συνεδρίου, πώς θα έχουμε έκθεση με βάση τις αποδόσεις και τις επιδόσεις στην ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα μας. Έχουμε και το κεφάλαιο 3 εστιάζουμε σε συγκεκριμένες πτυχές κάθε χρόνο. Υπάρχει και η δυνατότητα να έχουμε συνολική αναθεώρηση και επισκόπηση σε αιτήσια βάση. Όμως ήδη η δουλειά μας ε, έχει μπει στο αυλάκι και έχει δρομολογηθεί. Τώρα, ως προς τη συμμόρφωση υπάρχουν νομικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Στις αποδόσεις όμως και στην επί, στις επιδόσεις είναι διαφορετικό το θέμα γιατί έχει να κάνει με το σχεδιασμό της πολιτικής, με την εφαρμογή και ελοποίηση της υποπολιτικής, με την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της μεταρρύθμισης με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα κατά τη διαχείριση των διαφόρων προγραμμάτων, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή έχουν οργανωθεί οι υπηρεσίες και τα τμήματα για να έχουν συγκεκριμένα παραδοτέα και να καταλήξουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί αν διαβάσω τις εκθέσεις για την αποδοτικότητά μας που δημοσιεύαμε πριν από κάποια χρόνια, ουσιαστικά το κυρίως θέμα ήταν η συμμόρφωση. Τώρα όμως προσπαθούμε να ελέγξουμε το αναντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα. Και βεβαίως θα πρέπει η διαδικασία να ξεκινήσει από την αρχή και η Επιτροπή συνεχίζει να δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε για το πολιετές ε, ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, ότι δηλαδή υπάρχει προπολογισμό για την αποδοτικότητα. Αυτή αυτοί είναι στόχοι που μοιράζονται όλα τα θεσμικά όργανα και όντω είναι πάρα πολύ δύσκολο για πάρα πολλά χρόνια να ελέγξει κανείς τον προϋπολογισμό που δόθηκε για την ενίσχυση των επιδόσεων και είναι και δύσκολο να καθορίσει κανείς προπολογισμό ούτως ή άλλως συγκεκριμένο ή με αυτό το σκοπό την ενίσχυση των επιδόσεων. Όμως αποτελεί με βασικό μέλημά μας. τους ή άλλος συγκεκριμένο ή με αυτόν τον σκοπό την ενίσχυση των επιδόσεων. Όμως αποτελεί βασικό μέλημά μας. Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει άλλοι τέσσερις στο λόγο. Παρακαλώ η αλλω συγκεκριμενο η με αυτο Αγιάλα. Παρακαλώ. μελημα μα. ευχαριστω εχουν ζητησει αλλοι τέσσερι το λογο Σύντομα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Τομέ Μουγκουρούθα για την παρουσία του εδώ δεν ξέρω αν είναι τυχαίο βέβαια, ε, που ήταν ε, υπεύθυνο ε, για τις διοικητικές δαπάνες 11 με 15. Ε, εντάξει, αστείο είναι αυτό που είπα, φυσικά και δεν είχε κανένα περιθώριο λάθους και ενώ τώρα έχουμε 0,01 εν πάση περιπτώσει αστείο φυσικά αλλά ε, όσον αφορά τις ε, βοήθειες ε, που έχουν δοθεί σε διάφορες χώρες, ιδιαίτερως δε στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και εν πάση περιπτώσει μου φαίνεται σημαντικό επίσης που εστιάσατε στις εκθέσεις σχετικά με τις τι εκθέσει που κάνει δηλαδή το ελεγκτικό συνέδριο ε, και που εστιάζεστε ε, σε συγκεκριμένους ε, προβληματισμούς κυρίω όσον αφορά το κατά πόσον μπορεί να βρεθεί μια λύση για το υψηλό ποσοστό λάθος για, την, για τον ορίζοντα 2020 καθώς επίσης και για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη γιατί εδώ προκύπτουν πραγματικά μεγάλοι ε, κίνδυνοι ε, και ένα μικρό λάθος μπορεί να σημαίνει ε, π.χ. 40 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό και να μπορέσουμε να ελέγχουμε τέτοια προγράμματα όπου τα λάθη κοστίζουν πάρα πολύ. Επίσης, η εξέλιξη ε, ε, όσον αφορά τον έλεγχο μέσω της αποτελεσματικότητας. Ε, πιστεύετε ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι προετοιμασμένο έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτήν την επόμενη φάση που είναι και τόσο απαιτητική. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα για τα σχόλιά σας. Κοιτάξτε, εδώ ε, μου βάλατε παράσημα τα οποία δεν ε, ε, αξίζω, δηλαδή το θέμα των διοικητικών δαπανών εξαρτάται από τις ε, από τα διάφορα όργανα και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς συμβάλαμε μέσα από κατάλληλες σωστές συστάσεις για το θέμα αυτό ε, και όσον αφορά ε, και, την, και τη διαχείριση του δικού μας οργανισμού, του δικού μας σπιτιού κατά κάποιο τρόπο. Τα του οίκου μας έπρεπε να τα δούμε όσο και τα των άλλων. Επομένως δεν είναι δικά μου τα εύσημα μόνο. Όσον αφορά δε τα άλλα θέματα, να σας πω ότι η εμπειρία μου σε σχέση με την ε, έρευνα ε, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το ε, σώμα του οποίου προεδρεύω. Ασχοληθήκαμε με τις joint undertakings και όπως είπατε και εσείς εδώ έχουμε πραγματικά υψηλά ποσοστά σφάλματος. Το είπε εδώ και χρόνια αυτό το ελεγκτικό συνέδριο ότι το ποσοστό σφάλματος δεν εξαρτάται από την μεικτή ή την ε, ή την ε, αποκλειστική αρμοδιότητα αλλά εξαρτάται και από άλλα πολλά στοιχεία όταν, έχουμε, ε, ε, όταν απαιτείται η επεξήγηση κάποιων επενδύσεων, όταν απαιτούνται δικαιολογητικά για να καταβληθούν οι δαπάνες. Εκεί έχουμε μικρότερα περιθώρια ε, λάθους. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει ήδη κάνει μια έκθεση για την απλούστευση των διαδικασιών διερεύνησης Ε, σχετικά με ε, τις πληρωμές για τον ορίζοντα 2020 και τώρα θα ξεκινήσει ο έλεγχος ε, οι εκθέσεις για την απλούστευση έχει δεσμευτεί το ελεγκτικό συνέδριο ότι θα τις εφαρμόσει και σε άλλες περιπτώσεις όπως ας πούμε είναι η γεωργία ή άλλα εργαλεία. Τώρα, Κοιτάξτε, εγώ όταν έφτασα στο ελεκτικό συνέδριο, ξεκίνησα με μια, ε, ευθύνη, μια θέση η οποία ονομαζόταν έλεγχος της οικονομικής και νομισματικής κρίσης και όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε λοιπόν με τον τομέα αυτό συνειδητοποιήσαμε ότι ούτε το ελεγκτικό συνέδριο ούτε κανένας άλλος είχε τις, ε, τους πόρους ή τις ε, δομές σύμφωνα με την ε, τότε δομή που είχαμε ε, δεν είχαμε λέω την δυνατότητα να ασχοληθούμε με αυτό το νέο πεδίο το οποίο είχε μακροοικονομικά στοιχεία ιδιαίτερα έντονα είχε νομισματικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις που ξεπερνούσαν την παραδοσιακή δομή και αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε με διαφορετικό τρόπο. Θυμάμαι ότι κάναμε ε, μια εσωτερική έκκληση ε, των, ε, στους ελεγκτές του σώματος που είχαν, που είχαν εμπειρία. Ζητήσαμε την πραγματογνωμοσύνη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Μερικές φορές δεν προσλάβαμε και συγκεκριμένους συμβούλους για συγκεκριμένα θέματα έτσι ώστε ε, να δώσουμε οικονομική βοήθεια σε χώρες που την χρειαζόντουσαν, τεχνική αρρωγή στην περίπτωση και της ε, Ελλάδας, οικονομική ε, αρρωγή, δημιουργήσαμε το European Market Authority, την ΕΣΜΑ, Scrutiny Market Authority, αυτή είναι την αρχή εποπτείας της αγοράς η οποία θα ελεγχθεί άλλωστε σύντομα. Επίσης, ε, δημιουργήσαμε έλεγχο όλων των διαδικασιών ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα εντός το οποίο πρέπει να ε, εργαστούμε έχουμε στόχους συγκεκριμένους στόχους για το μέλλον. Θέλουμε να δουλέψουμε με βάση την ετήσια έκθεση και την ε, ε, αποτελεσματικότητα και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε και για να το επιτύχουμε βεβαίως χρειαζόμαστε ε, τεχνολογική προσαρμογή, χρειαζόμαστε τεχνικές όπως είναι τα big data ή τα open data χρειαζόμαστε χρήση καινοτομία. Πάντως πιστεύω ότι η νέα ευέλικτη δομή θα ε, επιφέρει οπωσδήποτε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και εγώ θέλω να ε, υποβάλω ε, ένα ερώτημα. Είναι μία στάνταρ ερώτηση. Πόσες μέρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο βρισκόσαστε στο Λουξεμβούργο. Έχετε κάποιο σπίτι, πηγαίνετε στο ξενοδοχείο. Okay. Well, time job. That's the eh. Η δουλειά μας ε, είναι πλήρους απασχόλησης. Αυτή είναι ε, η δουλειά μου, αυτό είναι το... Αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει. Ναι, έχω σπίτι στη... στο Λουξεμβούργο, αλλά έχω και σπίτι στην Μαδρίτη. Τα παιδιά μου σπουδάζουν εκεί αλλά τον περισσότερο χρόνο μου το περνάω στο Λουξεμβούργο. Και πολλά Σαββατοκύριακα πρέπει να σας πω, αλλά εντάξει αυτό το κάνω και όλος γιατί θέλω να γνωρίσω την περιοχή. Κοιτάξτε, η εντολή μας είναι να συμβάλλουμε ε, στην εργασία καθώς επίσης και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουμε συνεδριάσεις, συνεδριάσεις τομέων, ε, και θα μπορούσα ίσως να σας προτείνω όταν μας καλείτε εδώ ε, να μην, είναι, ε, να μην συμπίπτουν οι ημερομηνίε με τις συνεδριάσεις ε, που έχουμε εμείς στο ελεκτικό συνέδριο, γιατί σε αυτή την περίπτωση δυσκολευόμαστε. Και ενδεχομένως να έχασα κάτι στη μετάφραση γιατί δεν φορούσα τα ακουστικά μου. Ε, με μεγάλη μας ε, χαρά ακούσαμε ότι η προτεραιότητα είναι προφανώς να εργάζεται κανείς στο ελεκτικό συνέδριο. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Η μία είναι πολύ συγκεκριμένη, η άλλη γενικότερης φύσεως και θα ήθελα και η απάντηση να είναι αρκετά περιορισμένη. Είσαστε εισηγητής για τον έλεγχο που αφορά στα ευρωπαϊκά σχολεία. Πολύ συγκεκριμένη αυτή η ερώτηση. Σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην απαλλαγή το θέμα του ευρωπαϊκού ή των ευρωπαϊκών σχολείων. Και στο το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρει ότι το ελεγκτικό συνέδριο αντιμετωπίζει τα σχολεία με κάποια επιφυλακτικότητα. Και ρωτώ, εσεί πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και αν ναι πώ. Και η δεύτερη ερώτηση, επειδή εκπροσωπείτε τη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου στην Ισπανία αλλά και αλλού και προς άλλους ενδιαφερόμενου, ερωτώ, το ελεγκτικό συνέδριο αντιμετωπίζεται ω ε, εταίρο ή ω ένα ανώτερο όργανο το οποίο όλοι φοβούνται. Και ποιο είναι το όραμά σα, πώ θα θέλατε οι άλλοι να αντιμετωπίζουν το ελεγκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πρώτον, όσον αφορά στα ευρωπαϊκά σχολεία. Εδώ και πολλά χρόνια είμαι αρμόδιος ε, για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Έχουμε έναν ειδικό φορέα ε, που χρηματοδοτείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια ειδική μορφή διαχείρισης αυτού του φορέα. Και έχουμε διαπιστώσει ότι η διαχείριση υποφέρει. Το σύστημα δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Της διαχείρισης και γενικότερα το χρηματοοικονομικό. Εγώ είμαι απόλυτα σαφής σε αυτά που λέμε και συστήνουμε. Εγώ προσωπικά ε, παρουσίασα τα πορίσματά μας στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων όπου παρίστανται όλα τα κράτη-μέλη και τους έχω συστήσει να κάνουν κάτι και πράγματι ε, κάτι έκαναν τώρα έχουν νέα μορφή λογιστικών ε, νέα πλατφόρμα ηλεκτρονική νέα διαχειριστική δομή και ανεξάρτητα με το ε, πόσο καλή είναι στη διδασκαλία η κόρη μου παρακολούθησε ευρωπαϊκό σχολείο για κάποια χρόνια. Άσχετα από αυτό, εγώ αναφέρομαι σε θέματα οικονομικά, διαχειριστικά. Ελπίζω λοιπόν τώρα πλέον είναι περισσότερο σοβαρή και παρότι δεν είμαι πλέον αρμόδιος για τα σχολεία, ελπίζω να έχει γίνει κάποια πρόοδος εντωμεταξύ. Τώρα πώς μας αντιμετωπίζουν ε, οι υπόλοιποι φορείς. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ευρωπαϊκός φορέας και οποτεδήποτε ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ε, θεσμούς ή φορείς, τα κράτη-μέλη, προσπαθούμε να επιδεικνύουμε πνεύμα συνεργασία, να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με τους αρμόδιους, ε, με τους ομολόγους μας ε, στα κράτη-μέλη. Έχουμε οργανώσει μία συνάντηση για να εορτάσουμε την 400 η επέτειό μας και νομίζω ότι η συνεργασία με όλους τους ομολόγους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλή, αλλά βεβαίως και εμείς είμαστε υπόλογοι ε, στα κράτη-μέλη, παρουσιάζουμε τις εκθέσεις μας ε, στα κράτη-μέλη, στο Κοινοβούλιο, επίσης ε, στις εθνικές κυβερνήσεις και θέλω να πιστεύω ότι μας αντιμετωπίζουν ως ε, εταίρο, συνεργάτη που εργάζεται για το καλό όλων των ε, ενδιαφερομένων στην Ευρώπη. Παρακαλώ, κύριος Έρσπαχ. Οι εκθέσεις των ε, ελεγκτών θα πρέπει να είναι καθοριστική σημασία, να περιλαμβάνουν πολλέ πληροφορίε για, τα, για του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εκεί θα πρέπει να διαπιστώνουν την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων, της χρήσης κονδυλίων. Ε, όλα αυτά βασίζονται σε ε, θέματα συμμόρφωσης και αυτό ε, είναι πολύ περιορισμένο. Θα σας εξηγήσω ότι ακριβώς εννοώ ε, για το θέμα της ε, συμμόρφωσης. Ε, ως εκ τούτου, για το μέλλον, εμείς οι ευρωβουλευτές θα επιθυμούσαμε ένα έγγραφο το να περιλαμβάνει πολλές ε, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες για τις δαπάνες, το πώς αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των δαπανών. Χαίρομαι που μιλήσατε για έναν προϋπολογισμό που βασίζεται στην απόδοση, αλλά και όπως όλοι και άλλοι και εγώ ε, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό, τέθηκε προηγουμένως. Ποιοι είναι οι δείκτες απόδοσης, ποιος τους ορίζει, πώς ε, γίνονται μετρήσεις, πώς κάνετε τις συγκρίσεις. Εγώ προσωπικά Σχετικά με τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η προστιθέμενη αξία των δαπανών που επιφέρουν οι δαπάνες και πιο συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Μπορεί κανείς να κάνει μια σύγκριση και να πει ε, η Ευρώπη των 28 και οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέφεραν προστιθέμενη αξία σε κάτι που θα μπορούσε να κάνει ένα κράτος μέλος και πώς το παρουσιάζετε αυτό, πώς μπορείτε να έχετε ένα έγγραφο περισσότερο ενημερωτικό, περισσότερο ουσιαστικό που θα μπορεί και το Κοινοβούλιο να καταλάβει κατά πόσον πράγματι ε, μπορεί να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα στη χρήση των δαπανών. Συμφωνώ μαζί σας. Ο έλεγχος ως προς τη συμμόρφωση, αυτό είναι σημαντικό και είναι το σημαντικότερο όλων Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσον οι δαπάνες γίνονται με βάση την κείμενη νομοθεσία. Αν δεν ισχύει αυτό, ε, υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να αλλάξουν οι προτεραιότητες ο προπολογισμό με βάση την απόδοση. Αυτό ίσω είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή για όσου λαμβάνουν πολιτικέ αποφάσει. Για το ελεγκτικό συνέδριο, σημαντικό και έτσι θα συνεχίσουμε να πράττουμε. Μα ενδιαφέρει η ο έλεγχος της απόδοσης. Καλούμεθα να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ε, παρόλα αυτά θα είναι δική μας ευθύνη και στο μέλλον το θέμα της απόδοσης. Βεβαίως, η ενημέρωση για την απόδοση προϋποθέτει ενδελεχή ανάλυση, ε, σωστές προδιαγραφές και δείκτες και αυτό βεβαίως πάλι εξαρτάται από τη δική μας ε, την επαγγελματική κατάρτιση, αξιολόγηση, αλλά και από τους κανόνες. Σχετικά με την ευρωπαϊκή Προσθέμενη αξία, πράγματι αυτό είναι κέριο θέμα. Και το θέμα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμός και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ε, είναι προς όφελος όλων στην Ευρώπη. Αυτό πράγματι είναι μία πρόκληση. Ε, οφείλουμε να είμαστε παρόντες και όσο πιο φιδωλή είναι η πόρη και όσο λιγότεροι το χρηματοδοτούνται από τον προπλογισμό, τόσο πιο σημαντικό είναι και το πώς γίνεται η χρήση των κονδυλίων. Σαφήνεια λοιπόν στην παρουσίαση των εκθέσεών μας. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και νομίζουμε ότι πλέον ε, η παρουσίασή μας είναι πολύ καλύτερη. Εμείς είμαστε παρόντες και στο Twitter ε, προσπαθούμε να κοινοποιήσουμε τα πορίσματά μας. Έχουμε μία στρατηγική επικοινωνίας και δεν ξέρω κατά πόσον είναι πάντα εύκολο να είναι η γλώσσα μας πιο απλή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πράγματι όλα αυτά αποτελούν ένα πρόβλημα. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Τομέμου Κουρούθα για την παρουσίασή του. Κυρία Πρόεδρε, η διαδρομή του όντω είναι πραγματικά πολύ καλή και ως επιθερατής, επιθεωρητής οικονομικών και ως καθηγητής πανεπιστημίου. Ωστόσο, με ενδιαφέρει περισσότερο η θητεία του ως του ελεκτικού συνεδρίου. Ε, επιλέγει πρόεδρος του τμήματος 4 ε, του ελεγκτικού συνεδρίου από τους συναδέλφους του, από τους συναδέλφους του γιατί έλεγξε και έχει σημαντική διαδρομή στους ελέγχους. Έχει ελέγξει τις συμφωνίες ελευθερού εμπορίου με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία. Έχει ελέγξει ε, τα θέματα της μακροοικονομικής βοήθειας, των, ε, της στήριξης, όπως ε, της Ελλάδας για παράδειγμα, την, τα πεπραγμένα με τα rating agencies επίσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε το μέλλον. το ελεγκτικό συνέδριο πώς μπορεί να βοηθήσει για να προλάβουμε τέτοιες κρίσεις στο μέλλον. Οι πολίτες έχουν την εντύπωση ότι αυτή η οικονομική κρίση ε, ξεπεράστηκε επισήμως. Έχουμε όμως λαϊκιστικά κινήματα και τάσεις και απόψεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν πιστεί περί αυτού με τον έλεγχο των μέσων των εργαλείων, με τη δουλειά του ελεκτικού συνεδρίου. Πώς μπορείτε να συμβάλλετε για να προλάβουμε μελλοντικές οικονομικές κρίσεις τέτοιου είδους από τη στιγμή που έχετε αρμοδιότητα αλλά και εμπειρογνωμοσύνη αδιαφυσβήτητη με τους ελέγχους που έχετε διενεργήσει στο παρελθόν. Απάντηση. Κύριε Σαλαφράγκα, σας ευχαριστώ θερμά για την ερώτησή σας. Δεν είναι καθόλου εύκολη και χαίρομαι γι' αυτό. Προηγουμένως μιλούσα για την πρόκληση που αποτελούσε για το ελεγκτικό συνέδριο το καθήκον να κάνει τον έλεγχο των πραγμάτων που θεωρούνται θέματα οικονομικής, χρηματοπιστωτικής, δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Οι συστάσεις που έχουμε συντάξει μέχρι σήμερα θεωρώ ότι είναι εξατλητικές και συμβάλλουν στη βελτίωση τέτοιου είδους ε, σημαντικών διαδικασιών όπως είναι η οικονομική στήριξη, η τεχνική βοήθεια των χωρών σε κρίση, όπως είναι και τα απεπραγμένα και η διαχείριση και ο έλεγχος της διαχείρισης των διαφόρων οργανισμών και υπηρεσιών ε, οικονομικής και χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο, ξέρετε, της του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που δεν έχει κλείσει ακόμα, δεν έχει καν γραφτεί ακόμα στο σύνολό του. Είναι πράγματα εν εξελίξη, συζητώνται στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από πλευρά ελεκτικού συνεδρίου αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Κάθε δύο χρόνια παρουσιάζουμε το Landscape Review, επισκόπηση πεδίου, έτσι το ονομάζουμε, για τα ελλείμματα στις, ε, στους ελέγχους, accountability gaps, δηλαδή τα κενά στους ελέγχους. Και εκεί δείχνουμε ότι μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής δομής που προτείνεται για την οικονομική και χρηματοοικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση δεν εντάσσεται στο φυσιολογικό σύστημα της λογοδοσίας και της απόδοσης λογαριασμών. Έχω πολύ περιορισμένη εντολή, π.χ. στην Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε διοργανικούς θεσμούς όπως είναι ο ESM, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και δεν έχουμε αρμοδιότητα εκεί να τον ελέγξουμε ε, τα οικονομικά του πεπραγμένα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κλείσουν αυτά τα κενά στον έλεγχο το ελεγκτικό συνέδριο έχει ήδη ξεκινήσει να δουλεύει πάνω σε μια επισκόπηση πεδίου, landscape review, και θέλουμε να παρουσιάσουμε με συνεπή τρόπο όλα τα ευρήματά μας σε αυτό το τομέα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να δουλεύουμε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες συστάσεις. Πώς μπορεί δηλαδή ο έλεγχος να συμβάλλει περισσότερο στη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Εν συντομία να σας πω τα εξής. Η Επιτροπή μας αλλά και το Κοινοβούλιο ζητά ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Αυτό το στηρίζεται ή θεωρείτε ότι δεν, ε, δεν αρμόζει. Κοιτάξτε, οι εκθέσεις αναχώρα υπάρχουν. Εμείς δεν έχουμε την αρμοδιότητα να κάνουμε δήλωση για τη διαχείριση των κρατών μελών. Τα ανώτατα ελεγκτικά συνέδρια στα κράτη-μέλη το κάνουν αυτό. Θέλουμε εμείς να βοηθήσουμε όσους λαμβάνουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να πάρουν αποφάσεις πεφωτισμένες για προγράμματα που επηρεάζουν τα κράτη-μέλη. Γιατί βεβαίως τα προγράμματα τα τρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Υπάρχουν καλές πρακτικές, μη καλές πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές και νομίζω ότι τα έχουμε βελτιώσει πολύ. Έχουμε βελτιωθεί πολύ, είμαστε πολύ πιο διαφανείς στην έκθεσή μας, αυτό είναι σαφές. Έχουμε συχνό, συχνούς γύρους τραπέζης, ε, συχνή λογοδοσία με διαφάνεια παρουσιάζουμε τα ευρήματά μας. Βεβαίως έχουμε το error rate, τη συχνότητα ε, των σφαλμάτων. Έχουμε πολλές εκθέσεις που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και στη χώρα μου. Έχουμε πάντοτε συγκεκριμένα ευρήματα. Σύντομα στην Επιτροπή σας θα υποβάλω έκθεση για τη διαχείριση της βοήθειας στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένο αναχώρα σαν αντικείμενο θέμα έκθεσης από αυτό. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το σύστημα και σε σχέση με την ετήσια έκθεση. Η Επιτροπή έχει πολλές πληροφορίες και πολλά στοιχεία. Αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά των ανώτατων θεσμικών οργάνων που έχουν να κάνουν με τα κράτη-μέλη και με τα δικά τους συντάγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες και την ανταλλαγή απόψεων. Προχωρούμε με τον επόμενο υποψήφιο. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ich rufe auf die Anhörung ähm, κλείνει τη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 Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κυρίες και κύριοι, ε, είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι μεταξύ ε, που βρίσκομαι σήμερα εδώ ως υποψηφία από την Δανία για το ελεγκτικό συνέδριο. Πρέπει να πω ότι εγώ ασχολήθηκα με το θέμα του δημοσίου ελέγχου για πάρα πολλά χρόνια και ε, στην χώρα μου, τη Δανία, αλλά και σε άλλες ε, διεθνείς ε, θέσεις και οργανισμού. Κυρίως ασχολούμαι με έλεγχο και αναφορά συμμόρφωσης και αποδοτικότητας. Έχω συμμετάσχει σε έξι εκθέσεις, κυρίως όσον αφορά την βιώσιμη χρήση των πρώτων υλών, καθώς επίσης και για τους τομείς ασφάλειας και δικαιοσύνης έχω συμβάλει στη βελτιστοποίηση της διακυβέρνησης ε, του ελεκτικού ε, συνεδρίου, την ε, συνεχή κατάρτιση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου έτσι ώστε να ε, βελτιωθεί όσο γίνεται περισσότερο και να συμβάλλω στην καλή ε, απόδοση του ελεγκτικού συνεδρίου. Μαζί με τους ε, συναδέλφους μου έχουμε συμμετάσχει στην εκπόνηση εκθέσεων και στο δικό μου τμήμα αλλά και σε άλλα τμήματα ή στο σύνολο του ελεκτικού συνεδρίου και το κύριο μέλημά μου ήταν πάντα η ποιότητα και η σωστή αντιμετώπιση των εμπλεκομένων. Κατ' εμέ, ενεργή ε, συμμετοχή ε, είναι εκ των σε ένα συλλογικό σώμα. Ως ε, μέλος της Επιτροπής του, του ελέγχου των ικανοτήτων και απόδοση του προσωπικού θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σχέση μεταξύ των αναλόγων ελεγκτικών σωμάτων. Ε, εγώ επανειλημμένα έχω εκπροσωπήσει το ελεγκτικό συνέδριο ε, σε διάφορα φόρα, κυρίως ε, και από τη θέση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής των Επαγγελματικών Προσόντων. Θεωρώ ότι το ελληνικό συνέδριο πρέπει να είναι ε, ένα μερόληπτο ε, και ε, δεοντολογικά άρτιο όργανο και κατά αυτήν την έννοια και προς αυτήν την κατεύθυνση θα προσπαθήσω να βελτιώσω ακόμα περισσότερο την κατάσταση στο ελληνικό συνέδριο εάν επιβεβαιωθεί η θέση μου. Θα συνεχίσω ε, τους ελεγκτικούς μου, τον ελεγκτικό μου ε, ρόλο και τις, ελεγκτικός μου τις ελεγκτικές μου υποχρεώσεις με επαγγελματισμό και αντικειμενικότητα. Ε, θεωρώ ότι έφτασε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει στους πολίτες ότι μπορεί να αποτελέσει προστιθέμενη αξία και να βελτιώσει την ζωή τους. Ε, και, με τον, και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την προστασία ε, των συμφερόντων των Ευρωπαίων φορολογουμένων ε, και τον εντελεχή έλεγχο των δαπανών η συμμόρφωση και η απορρόφηση δεν μπορεί να είναι αρκετές διότι οι πολίτες θέλουν μετρήσιμα αποτελέσματα και επιτεύγματα. Κατά την έννοια αυτή, το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει και τη γνώση και την αντοχή και την ανθεκτικότητα να αντιμετωπίσει τους ε, κινδύνους. Όπως είπε και ένας καλός μου συνάδελφος, ε, θα πρέπει να προετοιμαστεί για το μέλλον ε, ε, ε, το, το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει και καλή συνεργασία ανάμεσα στο ελεγκτικό συνέδριο και τους πολιτικούς του εταίρους. Τα τελευταία χρόνια ήμουν στη διάθεση και της δικής σας Επιτροπής αλλά και άλλων Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με ε, κάλεσαν έτσι ώστε να αναφερθώ ενώπιον τους για την εργασία του ελεγκτικού συνεδρίου. γι' αυτό ζητώ την υποστήριξή σας για μια νέα εντολή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους σας για την προσοχή σας και έτοιμη να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις ε, που κάνατε, τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Έχω διαβάσει όλα τα έγγραφα και τις συνόψεις της καριέρας σας και των δραστηριοτήτων σας άκουσα και αυτά που μας είπατε μόλις τώρα. Και πραγματικά δεν έχω ερωτήσεις. Ε, εγώ έχω θετική άποψη σχετικά με την συνέχισή σας ε, εντός του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και καλύτερη ισορροπία φίλων στο ελεγκτικό συνέδριο δεν ε, σκεφτήκατε ποτέ ότι ίσως το, τα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου ε, θα πρέπει να ζητήσουν ίσως και από τα κράτη-μέλη περισσότερη ε, ισορροπία φύλων γιατί ίσως μέχρι το τέλος του Αρμαγεδόνος να μην έχουμε γυναίκες α, εκτός από τη Δανία, την Εστονία και τη Βουλγαρία. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε από κοινού έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η τόσο παλαιομοδίτικη στάση, η τόσο ξεπερασμένη στάση. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ κύριε Σεγητά για τα καλά σας λόγια. Όσον αφορά την ισότητα των φίλων στο ελληνικό συνέδριο, εσωτερικά πρέπει να σας πω ότι προσπαθούμε να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση έτσι ώστε να έχουμε σε ε, διηγητικές θέσεις ε, γυναίκες. γιατί αν θέλουμε να έχουμε ας πούμε διευθυντή γυναίκα θα πρέπει να έχουμε προηγουμένως φροντίσει στο προσωπικό να υπάρχει ισότητα ε, φίλων. Πρέπει να πω ότι έχω εκπλαγεί πολύ θετικά από το, ε, από το υψηλό επίπεδο ε, των του προσωπικού του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες και θέλουμε περισσότεροι auditing directors να είναι γυναίκες. όσον αφορά την ε, ισότητα φύλων, όσον αφορά τα μέλη του Ελεκτικού συνεδρίου. Έχουμε την Ουγγαρία, τη Γαλλία, τη Δανία και τη Βουλγαρία. Χαίρομαι ε, γιατί πριν από μερικές μέρες η Σουηδική κυβέρνηση ε, όρισε και μια νέα υποψήφιο γυναίκα για το Ελεκτικό συνέδριο. Θα φτάσουμε λοιπόν στον αριθμό των πέντε γυναικών στο Ελεκτικό συνέδριο. Ε, το οποίο είναι ήδη ένα καλό θέμα. Ε, και νομίζω ότι μόνο πιέζοντας διαρκώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, το επιθετικό αποτέλεσμα. Ναι, και εσείς από την πλευρά σας πιέζετε, πολύ ωραία. Είναι σημαντικό να ασκήσουμε πίεση από κοινού και προς πάσα κατεύθυνση. έτσι ώστε και στα διοικητικά συμβούλια γενικώ να έχουμε περισσότερε γυναίκε. Νομίζω ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση ακόμα περισσότερη. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ δύο ερωτήσεις που θέλω να υποβάλω προς όλα τα μέλη. Το θέμα της παρουσίας στο Λουξεμβουργό, αν έχετε κατοικία στο Λουξεμβούργο και κατά μέσο όρο πόσες ημέρες εργάζεστε στο ελεγκτικό συνέδριο. Και δεύτερον, οι συστάσεις αναχώρα, οι εκθέσεις αναχώρα. Αυτό το υποστηρίζετε ή όχι. Και αν ναι ή όχι, για ποιο λόγο. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που έκανα όταν με εκπλήξατε την προηγούμενη φορά που με υπερψηφίσατε, πήγα και νίκιασα διαμέρισμα στο Λουξεμβούργο. Εκεί ζω, είναι η μόνιμη μου κατοικια τέσσερι Τέσσερις-πέντε ημέρε την εβδομάδα εργάζομαι. Είμαι παρούσα δηλαδή στο ελεγκτικό συνέδριο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ που περπατάω κάθε πρωί και πάω στη δουλειά μου. Αυτό είναι ε, πολύ καλό, γιατί ειλικρινά σα λέω και στο Λουξεμβούργο έχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση ε, ημέρε. Ε, στις, ε, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Κατά τα άλλα, Σχετικά με τις εκθέσεις αναχώρα γνωρίζω ότι έχετε δείξει το θέμα αυτό ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρξουν και άλλες αναλύσεις, δηλαδή κάποιες ε, ειδικέ εκθέσεις για κάποιες συγκεκριμένες χώρες ή ε, περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένες χώρες να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Νομίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο έχει προχωρήσει πάρα πολύ για να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες για κάποιες χώρες και να τις εντάσει στην ετήσια έκθεσή του. Προς εκεί βαδίζουμε, δεν έχουμε επιτύχει ακόμα το στόχο μας. Όσον αφορά τις ειδικέ εκθέσεις, νομίζω ότι έχουμε ε, ένα πολύ καλό μείγμα διαφόρων προγραμμάτων σε διάφορες χώρες και Νομίζω ότι μπορούμε πράγματι να εστιάσουμε σε μία χώρα. Νομίζω όμως ότι για έναν ελεγκτή αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αν επιλέξει περισσότερες χώρες μπορεί να κάνει τη σύγκριση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Για μένα λοιπόν ε, το να ελέγχουμε μία και μόνο χώρα, ίσως αυτό να μην είναι τόσο αποτελεσματικό, γιατί δεν έχει κανείς ε, το κριτήριο της σύγκρισης και δεν μπορεί, όπως σας είπα, να συγκρίνει με άλλα κράτη-μέλη. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο συνάδελφος κύριος Τάραντ. Βεβαίως χαιρόμαστε διότι είστε γυναίκα και μέλος του ελεκτικού συνεδρίου και μάλιστα ε, με ακτιβισμό και επαγγελματισμό προσπαθείτε να καταφέρετε να είναι περισσότερες οι γυναίκες στις ε, υψηλές θέσεις διοίκησης, στις ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας του ελεκτικού συνεδρίου. Το επάγγελμα άλλωστε του ελεγκτή δεν ε, ήταν γυναικοκρατούμενο επάγγελμα και γι' αυτό το ότι υπάρχετε και η παρουσία σας εκεί είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας. Από εκεί και πέρα, έχετε μεγάλη εμπειρία στο διεθνές στερέωμα και γνωρίζετε, το λέτε κι εσείς, ότι εμείς έχουμε πρόβλημα με τα καταπιστευματικά ταμεία, τα οποία όλο και περισσότερο θα πολλαπλασιάζονται και μας φαίνεται αυτό πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και άλλες ε, λύσεις και ποια είναι η λύση κατά τη γνώμη σας ε, για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο, πώς θα κυκλοφορεί με τον καλύτερο τρόπο με εντό καταπιστευματικού ταμείου τα χρήματα που θα κυκλοφορούν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα πρέπει όλα αυτά να εμφανίζονται στον προϋπολογισμό. Και από τη στιγμή που και εσείς είστε ελεγκτής προσωπικά και έχετε ασχοληθεί με την ε, με τα εσωτερικά του ελεγκτικού συνεδρίου σε επίπεδο προσωπικού στο ελεγκτικό συνέδριο. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να έχουμε πραγματικό έλεγχο του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Έχουμε αρκετό υλικό, έχουμε καλά προετοιμάσει τους ελεγκτές για να περάσουμε σε προϋπολογισμό και έλεγχο του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις απάντηση. Σας ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ για το ερώτημα. Το πρώτο σας ερώτημα για τα καταπιστευματικά ταμεία ε, είναι ενδιαφέρον και θα ήθελα να πω ως προς το θέμα αυτό ότι η έκθεση ήταν ε, σημαντική για το πρώτο καταπιστευματικό ταμείο το οποίο εξετάσαμε, το πρώτο Trust Fund. Μεγάλο μέρος της στήριξης δίδεται με τη μορφή της στήριξης στον προϋπολογισμό και έτσι ένας ελεγκτής δυσκολεύεται να ακολουθήσει τη ροή του χρήματος. Είναι σαν να αναμειγνύει κανείς το ζεστό με το κρύο νερό και είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς που ακριβώς πηγαίνει μέρος των χρημάτων ξεχωριστά. Το σημαντικό είναι ότι Χρειαζόμαστε σαφείς στόχους από πλευράς ε, Επιτροπής, σαφείς επιδιώξεις και σαφείς δείκτες. Όχι πολλούς, γιατί νομίζω ότι η Επιτροπή δυσκολεύεται να μας δώσει αρκετά μεγάλο αριθμό στόχων και δικτών. Όμως χρειαζόμαστε τους σωστούς δείκτες, τους σωστούς στόχους, αυτά που θα μας στείλουν προς τη σωστή κατεύθυνση για να έχουμε σωστή επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αντίκτυπο στους αποδέκτες τους. Και πιστεύω ότι εάν ε, δούμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα δούμε ότι η στήριξη δίδεται με πολλούς και διαφορετικούς ε, τρόπους. Έχουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, έχουμε τα καταπιστευματικά ταμεία, την άμεση στήριξη, με διάφορα κανάλια. Με διάφορους διάβλους δίδεται η βοήθεια ή η στήριξη. Ως ελεκτής όμως, εγώ θέλω διαβεβαιώσεις ότι τα χρήματα δαπανήθηκαν σωστά και ότι παρήχαν τους πόρους και οδήγησαν στα αποτελέσματα που επιθυμούσαμε, γιατί οι φορολογούμενοι αυτό θέλουν να γνωρίζουν, ότι η βοήθειά μας πράγματι στηρίζει τον κόσμο και τους ανθρώπους και τους λαούς στην οποία, στους οποίους τη δίνουμε αυτή τη βοήθεια. Αυτό που λέτε χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες και ως ελεγκτές πρέπει να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος να ακολουθούμε τη ροή του χρήματος, να ακολουθούμε το χρήμα και να δούμε πώς θα μετρήσουμε τον αντίκτυπο που έχει αυτή η στήριξη. Τώρα για τα οργανωτικά του ελεγκτικού συνεδρίου, αν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό. Πολύ εύκολο είναι να πω ναι προσλάβετε κι άλλους, δώστε μας κι άλλο προσωπικό. Πάντοτε θα μας χρειάζεται και πάντοτε θα το θέλουμε, αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Πιστεύω ότι σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον ελέγχου πρέπει μονίμως να είμαστε βέβαιοι ότι ενημερώνουμε ε, την επιστημονική μας γνώση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο να μπορούμε να έχουμε προϋπολογισμό με βάση τις επιδόσεις και την απόδοση και τα αποτελέσματα, όμως πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε αυτό το τομέα της επιμόρφωσης και της συνεχούς αναβάθμισης και ενημέρωσης επικαιροποίησης ε, των ε, γνώσεών μας. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Λαμπάγιοβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ποιοι έλεγχη συγκεκριμένη με θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη θα θέλατε να δημιουργήσετε ή να προωθήσετε ή να θεσπίσετε. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ενδιαφέρουσα και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι η έκθεσή μου για τα απορρίμματα τροφίμων, food waste, ήταν μια έκθεση που έδειχνε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο τις υφιστάμενες πολιτικές. Δεν ζητούμε επιπρόσθετη χρηματοδότηση, αλλά επιδιώκουμε να ε, αξιοποιήσουμε καλύτερα τις υφιστάμενες πολιτικές και με αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Ξέρετε, ποτέ δεν είχαμε τόσα ανακοινοθέντα τύπου και δελτία τύπου ε, όσο για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήρθε σε μια πολύ κατάλληλη χρονική στιγμή ε, να συμπέσει η έκθεσή μας με την ε, δημοσίευση της δικής σας έκθεσης στη δική σας επιτροπή και έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στη δική σας δουλειά. Και να είναι στραμμένο το ενδιαφέρον μας στους πολίτες. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών που έχουμε δημοσιεύσει για το 2018 περιλαμβάνουν διάφορες εκθέσεις για τα θέματα αυτά, για τα βιολογικά τρόφιμα, για τα δικαιώματα των επιβατών, για την ανεργία των νέων. Νομίζω ότι αυτές οι εκθέσεις πραγματικά είναι άριστα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο το ελεκτικό συνέδριο δείχνει ότι συντάσσει εκθέσεις για θέματα που αφορούν τον Ευρωπαίο πολίτη πραγματικά και ε, μπορεί να βοηθήσει την ε, δουλειά της δικής σας Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και για μας βέβαια αυτή η έκθεση για το καταπαστευματικό ταμείο, γενικά για τα καταπαστευματικά ταμεία ήταν πολύ σημαντική και μας, με χαρά ακούσαμε ότι ε, πολλές φορές τα, οι διαχειριστικές δαπάνες καταβάλλονται και δύο και τρεις φορές. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Αναφερθήκατε στην βοήθεια στον προπολογισμό. Αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και είπατε ότι θέλετε να μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι πράγματι τα χρήματα ε, καταλήγουν ε, εκεί για το οποίο είχαν ε, προβλεφθεί. Αυτό όμως σε, αυτό το, αυτή τη βοήθεια, σε αυτό το επίδομα δεν μπορεί κανείς να το ισχυριστεί. Βέβαια από την άλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίζεται με μανία μάλιστα αυτό το θέμα και για μένα δεν είναι απόλυτα κατανοητό. Θα ήθελα να γνωρίζω Πώς ακριβώς είναι η συνεργασία σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις εκθέσεις ε, δεν μπορεί κανείς να δει ε, κατά πόσον η Κομισιόν ε, δέχεται τις προτάσεις σας ή όχι. Και θέλω να ερωτήσω, εκεί που εκεί έλεγχοι, εσείς μεταβαίνετε εκεί προσωπικά, γιατί πολλές φορές ε, βλέπουμε ότι η Κομισιόν ε, πηγαίνει και επισκέπτεται τόπου μόνο τα σημεία εκείνα που όλα λειτουργούν μια χαρά και αποφεύγει να επισκεφτεί τους τόπους και χώρους όπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Όσον αφορά το καταπίστευμα, θέλω να σας πω ότι η σύστασή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ότι θα έπρεπε να ε, πάρουμε ε, τις συστάσεις από αυτό το καταπίστευμα να τις εντάξουμε σε άλλα τα οποία έχουμε προβλέψει για το μέλλον και υπάρχουν πολλά θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τα μελλοντικά καταπιστεύματα αν ε, θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο χρηματοδότησης. Και όσον αφορά στην ερώτησή σας για το κατά πόσον ε, θα πρέπει να επισκεπτόμεθα χώρες ή όχι, δηλαδή ή αν προτιμάμε να πηγαίνουμε σε χώρες εκεί που τα πράγματα λειτουργούν μια χαρά. Θέλω να σας πω ότι εμείς όταν κάνουμε τους ελέγχους μας ε, πάντα κάνουμε αξιολόγηση κινδύνου και έχουμε ένα μεγάλο μείγμα ελέγχων όπου γνωρίζουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα, θα δώσουμε καλά παραδείγματα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου γνωρίζουμε ότι εκεί πρέπει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις και ότι ε, πρέπει να ε, υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Αυτή η έκθεση για το ε, ταμείο για το οποίο συζητάμε θα συνεχίσουμε να ζητάμε νέες πρωτοβουλίες για να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία μας και αυτή να καταλήξει σε νέες πρωτοβουλίες που ενδεχομένω αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση σας. Πολύ ωραία. Ε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και χαιρόμαστε για τη μελλοντική μας συνεργασία. Και τώρα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 welcome to the committee. And you get immediately the floor. You get immediately the floor to present. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Έχετε αμέσως το λόγο για να μας παρουσιάσετε την ομιλία σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο για αυτήν την ε, αρχική παρέμβαση. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, χαίρομαι που βρίσκομαι για μία ακόμα φορά ενώπιόν σας ως ε, υποψήφιος ε, ε, ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου μετά από αίτημα σχετικό των αρχών της χώρας μου. Πριν από ένα χρόνο παρουσιάστηκα ενώπιόν σας έτσι ώστε να μου δώσετε την θετική σας γνώμη για να συνεχίσω στην θητεία του προκατόχου μου Πορτογάλου μέλους του ελεγκτικού ε, συνεδρίου. Έχω υποβάλει και μια σύνθεση, μια σύνοψη όπως μου ζητήθηκε καθώς επίσης και αναλυτικό βιογραφικό μου σημείωμα. Έχετε λοιπόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το παρελθόν και είμαι στη διάθεσή σας να σας υποβάλω οποιασδήποτε επιπλέον ε, πληροφορίες μου ζητήσετε. Αλλά το σημαντικό είναι να μιλήσουμε τώρα για το παρόν και για το μέλλον. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ε, είμαι απολύτως δεσμευμένος στον ρόλο που οφείλει να παίξει το ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά την διαχείριση του κόστους και τον έλεγχο των δαπανών, έτσι όπως αναφέρεται σε τις ε, συνθήκες. Ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εμπιστεύονται τους διαχειριστές των ε, χρημάτων τους. Γι' αυτό λοιπόν αποδίδω ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου καθώς επίσης ε, και την δήλωση συμμόρφωσης όσον αφορά τις δαπάνες. Τα δύο αυτά ε, έγγραφα έχουν συμβάλει ε, στην ε, βελτίωση της, της υγιούς οικονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπωσδήποτε η προσέγγιση θα πρέπει να είναι διαρκώς εξελισσόμενη, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία των άλλων ελεγκτών, έτσι ώστε σιγά σιγά να μειωθεί η ανάγκη ελέγχου των ευρωπαϊκών ενωσιακών οικονομικών. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται βεβαίως υπό το κράτος δικαίου, αλλά θα ήθελα στα επόμενα χρόνια να αυξήσουμε την εστίασή μας σε συγκεκριμένα ζητήματα, ε, ε, μετρήσιμα αποτελέσματα ε, και μετρήσιμη αντιμετώπιση των αντικτύπων που οι αποφάσεις μας μπορεί να έχουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να προοδεύσουμε ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά ε, είναι άλλωστε στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο στρατηγικό έγγραφο του ελεγκτικού συνεδρίου το οποίο και εγώ ίδιος έχω προσυπογράψει και το οποίο με δεσμεύει απολύτως. Επίσης να σας πω ότι ε, είμαι τώρα υπεύθυνος ε, του τμήματος δαπανών του ελεγκτικού συνεδρίου. Γνωρίζω ότι η νέα δημοσιονομική περίοδος ε, και επομένως το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να συμβάλλει ε, μέσω της ανάλυσης ε, του ισχύοντος δημοσιονομικού ε, πλαισίου κυρίως λαμβάνοντας υπόψη την ε, γεωργία ε, της οποίας το οικονομικό βάρος ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νέοι δημοσιονομικοί περιορισμοί θα προκύψουν και επομένως προκύπτει, προκύπτουν νέες ανάγκες όσον αφορά τις ενωσιακές και δημόσιες πολιτικές. Επίσης, νέες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, την άμυνα και την ε, μετανάστευση, καθώς επίσης ε, ε, πολύ σημαντικό θεωρώ και τον κλάδο του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Πολλές είναι οι προκλήσεις τις οποίες γνωρίζετε και εσείς. Όπως είπα και ένα χρόνο πριν στην Επιτροπή σας, εγώ πιστεύω ότι αποτελεσματικά θα μπορέσουν όλοι να αντιμετωπίσουν το διακύβευμα, την πρόκληση αυτή μονάχα εάν παραμείνουν, εάν παραμείνουμε ενωμένοι. θεωρώ και το έχω πει επανειλημμένα και το επαναλαμβάνω εδώ ότι το ελεγκτικό συνέδριο χρειάζεται ανεμεροληψία και ανεξαρτησία. Ε, αυτά άλλωστε αποτέλεσαν και τα βασικά στοιχεία τα οποία με οδήγησαν και στην προηγούμενη ε, καριέρα μου και στις προηγούμενες ε, θέσεις μου. Θεωρώ ότι ο καλός διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εκ των ουκάνευ ιδιαίτερος φύσεως της με αυτήν την Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριε συγητά με τούτη την παρέμβασή μου ελπίζω να ε, σας έπεισα ε, για την ε, καλή συμμετοχή μου στις εργασίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα περιμένω με μεγάλη προσοχή σχόλια και παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντεφιγκορέιντο, Έχω δύο ερωτήσεις που αφορούν στις δραστηριότητες σας ε, ως ε, ελεγκτής για θέματα κοινή γεωργικής πολιτικής. Πιστεύετε ότι το να κάνει κανείς έναν έλεγχο και το να προσπαθεί να διαπιστώσει ενδεχομένως ε, κατά πόσον κάποιες επιδοτήσεις ε, ε, δημιουργούν, προκαλούν ανισότητες ανάμεσα στα παλαιότερα και τα νεότερα κρατημέλη. Μήπως υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία, συμφωνείτε από αυτού. Και δεύτερον, πιστεύετε ότι ήταν χρήσιμο το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει έναν σωστό έλεγχο πριν από την ψηφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα ζυζανιοκτώνων και λοιπασμάτων. Αυτές τις δύο ερωτήσεις είχα να σας υποβάλω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάραντ για τις ε, ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα εξ αυτών είναι το εξής. Κατά πόσον οι επιδοτήσεις ε, που χορηγούνται στο πλαίσιο της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής, κατά πόσον είναι αποτελεσματικές ή όχι, αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, υποβάλλεται μία ερώτηση που αφορά στην ισότητα Όσον αφορά το πρώτο θέμα, εγώ θα ήθελα να πω από αυτό το εξή. Πιστεύω ότι όλοι οι μηχανισμοί, οι οικονομικοί, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής και έχω κατά νου τη μεταρρύθμιση που ετέθησε ισχύ το 2015 και τα νέα προγράμματα πληρωμών, καταβολής επιδομάτων στους γεωργούς. Έχοντας λοιπόν αυτά κατά νου, θα ήθελα να πω ότι πράγματι διαπιστώσαμε ότι στην αρχή υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Αλλά οι μηχανισμοί χρηματοδότησης Γενικότερα ε, λειτουργούν εύρυθμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας πιστεύουμε ότι τα προβλήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο για πολλά κράτη-μέλη να θέσουν σε ισχύ αυτούς τους ε, μηχανισμούς μεταρρύθμισης. που αποφασίστηκε το 2015. Βέβαια, τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά, με κάποιες δυσκολίες και κάποια προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι λειτουργούν καλά. Και αυτός ε, είναι ένας από τους λόγους γιατί στο, στην έκθεσή μας, το κεφάλαιο που έχει σχέση με τους ε, φυσικούς πόρους, εκεί αναφέρουμε ότι πράγματι υπάρχει μικρότερο ποσοστό σφαλμάτων. Δεύτερη ερώτηση. Αυτή που έχει σχέση με το περιβάλλον και τη στάση έναντι αυτού. το δούμε αλλιώ. Ας πάρουμε το θέμα της γεωργικής πολιτικής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Εμείς θεωρούμε ότι με τη μεταρρύθμιση του 2015 ο νομοθέτης είχε κατά νου στη γεωρική πολιτική να εντάξει και κάποια στοιχεία που έδειχναν ότι ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον. Υπάρχει αυτό στους κανονισμούς. Όμως, παρά τις καλές προθέσεις, τελικά αυτά όλα δεν οδήγησαν σε αλλαγή της συμπεριφοράς των γεωργών. Δηλαδή, καλές ήταν οι προθέσεις, αλλά δεν υπήρχαν ε, αρκετοί επαρκανοποιητικοί μηχανισμοί για να επιφέρουν τα ευκταία αποτελέσματα που ήταν η προστασία του περιβάλλοντος. Από ό,τι φαίνεται, στο μέλλον αυτό ο νομοθέτης ε, πρέπει να το λάβει υπόψη του. Σε κάτι άλλο θα αναφερθώ. Ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε τη μεταρρύθμιση του, το 2015 αλλά και το 2009 Ένα από του λόγους ήταν να υπάρχει ισότητα. Ισότητα ανάμεσα στους γεωργού γεωργούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και πιστεύουμε ότι έγιναν κάποια σωστά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε όμως ότι ε, προ αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνουν και πολλά άλλα. Ε, δεν ξέρω αν απάντησα ικανοποιητικά στι ερωτήσει σα. Ναι, ε, περι... περιμένουμε την ειδική έκθεση. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much. Uh... Για το πρασίνισμα. Ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα για την... Ποια είναι κατά την άποψή σας η μεγαλύτερη αδυναμία στο τρόπο με, στη διαδικασία με την οποία επιτολεί το έργο του το ελεκτικό συνέδριο. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Εγώ Μόνο ένα χρόνο βρίσκομαι στο ελεγκτικό συνέδριο και δεν είναι εύκολο για μένα να μιλώ για τις αδυναμίες. Πιο εύκολα μπορώ να μιλήσω για τα θετικά στοιχεία, κυρίως για τους ανθρώπινους πόρους. Βρήκα εξαιρετικό προσωπικό, ε, ανθρώπους εξαιρετικά καταρτισμένους, πολύ καλούς επαγγελματίες, με μεγάλο κίνητρο. Είναι εξαιρετικό να μπορεί κανείς να συνεργάζεται με τέτοιους ανθρώπους. Τώρα, ποια είναι τα τροτά σημεία και οι αδυναμίες. Από τη σύντομη θητεία μου μέχρι σήμερα, κάτι που είδα είναι ότι είναι δύσκολο να είναι πραγματικά αποτελεσματική η συνεργασία μεταξύ του ελεκτικού συνεδρίου και των ανώτατων εθνικών κρατικών ελεγκτικών αρχών, δηλαδή αντιστοίχων ελεγκτικών συνεδρίων. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα γιατί βεβαίω είμαστε ανεξάρτητες οντότητε. Θα πρέπει όμως όλοι να γνωρίζουν ότι εμείς έχουμε την αρμοδιότητα του εξωτερικού ελέγχου των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των εθνικών πόρων και ευρωπαϊκών πόρων και ότι θα έπρεπε να βρούμε και ότι πρέπει να βρούμε μηχανισμού συνεργασίας και συντονισμού των δραστηριοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν τα καταφέρουμε, αυτό θα είναι πολύ καλό αποτέλεσμα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα μειωθούν οι έλεγχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μειωθεί και το διοικητικό βάρος, το διοικητικό άχθος, το οποίο αναφέρθηκα στην αρχική μου δήλωση. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το βασικό ζήτημα, πώς θα διασφαλίσουμε δηλαδή ότι στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καλή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ του ευρωπαϊκού επίπεδου ελέγχων και των εθνικών. Ευχαριστώ. Ε, Ακούσαμε και τις ε, τεγκόμοι για τους συνεργάτες του Ελληνικού Συνεδρίου, παρότι σε εμά ε, στη Γερμανία λέμε ότι και πολλοί έπαινοι είναι περιττοί. Ο κύριος Αλαφράγκα. Σας ευχαριστώ κύριε Φικέη Ρέντο για την παρουσίασή σας. Διάβασα με μεγάλη προσοχή το βιογραφικό σας σημείωμα. Ε, αντιλήφθηκα την ευρία εμπειρία που έχετε στην Πορτογαλία στο θέμα των ελέγχων και είδα και τις εκθέσεις που έχετε υπογράψει κατά τη θητεία σα ω μέλος στο ελεγκτικό συνέδριο. Στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική, από ό,τι, καταλαβαίνω, εσείς, ε, ε, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς αποτελείτε μέρο της Επιτροπής Διαοντολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν θέλω βεβαίω να σας θέσω αδιάκριτες ερωτήσεις για υποθέσεις και φακέλους που είναι εμπιστευτικοί και με τους οποίους ασχολείται η Επιτροπή δεντολογία στην οποία παρίσταστε. Θα ήθελα όμως να μας υπενθυμίσετε ποιε είναι οι δραστηριότητε που είναι συμβατές με ε, το θεσμικό όργανο. Δηλαδή δεν θέλουμε να μας πείτε συγκεκριμένα πρόσωπα, νούμερα και αριθμούς, αλλά ε, να μας πείτε το πεδίο αρμοδιοτήτων. Ευχαριστώ. Απάντηση. Κύριε Σαλαφράγκα, σας ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα, για το ερώτημα. Μία είναι η ερώτηση που μου αμπευθύνεται Και σας ευχαριστώ που διαβάσατε και τις εκθέσεις ε, για τις οποίες είχατε την ευθύνη στο πλαίσιο του ελεγκτικού συνεδρίου. Αναφορικά με το ερώτημά σας, δεν δυσκολεύομαι να απαντήσω, γιατί υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας και για τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου και για το προσωπικό, το διοικητικό. Και αυτός ο, ο κώδικας δεοντολογίας εκφράζει όλες τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται, που πρέπει να εφαρμόζονται στην ε, δημόσια διοίκηση. Μιλούμε για ακαιρεότητα, αμεροληψία, ανεξαρτησία, συναδελφικότητα. Αυτά, αυτές είναι οι βασικές αξίες και όταν έχουμε περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας, προσπαθούμε Προσπαθούμε πάντοτε να εφαρμόζουμε τους γενικούς κανόνες στα διάφορα διεθνή ε, κείμενα που υπάρχουν και στις διάφορες συνθήκες και αυτά τα συμπεριλαμβάνουμε, τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Για παράδειγμα, ε, έχουμε άλλες δραστηριότητες που ενδεχομένω μέλη θέλουν να εφαρμόσουν εκτός ελεγκτικού συνεδρίου. Νέες δραστηριότητες ε, με τις οποίες θέλουν να ασχοληθούν τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου μετά το τέλος της θητείας τους. Όλα αυτά είναι περίπλοκα ζητήματα. Υπάρχουν ερωτήματα με τη συμμετοχή σε ορισμένους ελέγχους διότι ενδεχομένως μπορεί να συνδέονται με προηγούμενες θέσεις και επαγγελματικές, ε, ε, επαγγελματικές θέσεις στη στρατιδιοδρομία του μέλους ή του ελεγκτή. Η Επιτροπή λοιπόν Οδοντολογίας ασχολείται και με αυτά και με τα διάφορα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Εθνών, ε, του ΩΣΑ, αλλά και βεβαίως και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν επίσης κανόνες. Όταν έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, πρέπει να γνωρίζουμε όλους αυτούς τους κανόνες και να ε, τους ε, ε, λάβουμε υπόψη και να βρούμε την καλύτερη λύση για την εκάστοτε υπόθεση. Δεν ξέρω αν σας απάντησα. Εάν όχι, ευχαρίστως να επεκταθώ περαιτέρω. συνάδελφος Έρσουαστ στον κατάλογο των ομιλητών. Κύριε Φιγκουρέντο, ως ε, ελεγκτής ε, σας ε, καλώ να ελέγξετε και τον εαυτό σας. στο ερωτηματολόγιο τίθενται ερωτήματα, ποια είναι τα του και οι αδυναμίες του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά θέλω να αξιολογήσετε εσείς τον εαυτό σας και να μας πείτε ποια είναι τα υπέρ και τα κατά σας. Η βασική μου αδυναμία είναι ότι δεν ξέρω τίποτα. Ότι πρέπει να μάθω πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου στο ελεγκτικό συνέδριο με όλη μου την καρδιά, γιατί εκείνοι έχουν γνώση που δεν διαθέτω εγώ. Και εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάνω σωστά τα μαθήματά μου σε εισαγωγικά, αν τους ακούω βέβαια και σωστά, αν ακούω αυτά που λένε οι συναδελφοί μου. Ξέρετε, αυτή είναι η προσέγγιση μου, αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Και φαντάζομαι με ρωτήσατε για αδυναμίες ε, στην επαγγελματική μου ζωή και όχι στην ιδιωτική μου ζωή, γιατί στην ιδιωτική μου εκεί και να δείτε αδυναμίες που έχω, αλλά δεν φαντα... μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα σας ενδιαφέρουν. Ναι, εντάξει, μπορεί να παίζουν ρόλο και οι αδυναμίες στην ε, προσωπική ζωή, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο σημαντικές. Όσον αφορά τώρα, αυτά για τις αδυναμίες μου και τώρα για τις ε, θετικές μου, θετική πλευρά του εαυτού μου είναι στα διαδρομία μου. 30 χρόνια στα διαδρομία σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης στην Πορτογαλία, σε πάρα πολλούς ε, τομείς ε, συνεργάστηκα με την εκτελεστική, την νομοθετική, τη δικαστική εξουσία. Είμαι μέλος ε, της κυβέρνησης στην ε, Πορτογαλία σε ανώτερους θεσμούς. Έχω εργαστεί στην Πορτογαλία, αλλά όχι μόνο. Έχω εργαστεί και στην Κίνα και σε άλλους ε, διεθνείς οργανισμούς ως εμπειρογνώμων. Νομίζω αυτό είναι το θετικό στοιχείο του εαυτού μου και κάθε μέρα προσπαθώ να δώσω και το καλύτερο. Αν το κάνω αυτό όλοι θα είμαστε σε σωστό δρόμο. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, όπως ρωτάω και όλους τους άλλους ε, που θέλουν την παράταση, αν μένουν στο Λουξεμβούργο, αν έχουν ε, κατοικία στο Λουξεμβούργο και ποια είναι η στάση τους για τις συστάσεις αναχώρα. Εκθέσεις μάλλον αναχώρα. Κυρία Πρόεδρε, η πρώτη απάντηση είναι ναι. Και εγώ, κατοικία, η μόνη μου κατοικία μου είναι στο Λουξεμβούργο. 30 λεπτά, μισή ώρα περπατάω, ε, πάω στο ελεγκτικό συνέδριο. Μ' αρέσει πολύ το Λουξεμβούργο, το χαίρομαι πολύ που είμαι εκεί. Και η δεύτερη ερώτησή μου έχει σχέση με τον ένα λιγάκι θαραλέος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ονοματίζει χώρες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ανάμεσα ε, στους θεσμούς, στις σχέσεις ε, θεσμών με τους πολίτες. Ε, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα στο να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα όπως το κάναμε φέτος αν αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε τις καλές πρακτικές ή για να πούμε ότι δεν υπάρχουν καλές πρακτικές στην ΑΒ χώρα. Υπάρχουν καλές πρακτικές και υπάρχουν και κακές πρακτικές σε όλες τις χώρες. Και το έχω δει αυτό με τα μάτια μου στην κοινή γεωργική πολιτική. Βλέπω να υπάρχουν καλές πρακτικές σε όλες τις χώρες και βλέπω ε, κακά παραδείγματα σε όλες τις χώρες, πάλι σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Νομίζω ότι είναι καλό το να υπάρχει διαφάνεια, να λέει κανείς ε, τα πράγματα με το όνομά τους και αν το κάνουμε αυτό ε, με στόχο να έχουμε καλύτερες οικονομικές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το πιο σωστό σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτός είναι ο στόχος, τότε νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε και γι' αυτό. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και η κυρία Γιάλα είναι η τελευταία που θα κάνει ερώτηση. Παρακαλώ. Με κάλυψε ο κύριος Αλαφράγκα για να είμαι ειλικρινής. Ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω ε, για την παρουσία σας στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για τα στατιστικά, γιατί ασχολείστε με πάρα πολλές περιπτώσεις ε, που έχουν να κάνουν με σύγκρουση συμφερόντων ή με θέματα που μπορούν να πλήξουν τη φήμη και το κύρος του ελεγκτικού συνεδρίου. Άλλωστε είστε μέλη ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου που ε, έχει να κάνει με όλα τα κράτη-μέλη. Από στατιστική σκοπιά η δουλειά της Επιτροπής Δεντολογίας είναι πολύ. Δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει θέμα δεοντολογίας. Και πώς συζητάτε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη φήμη του ελεκτικού συνεδρίου και την προστασία του κύρους του. Αυτό καταρχάς, κατά δεύτερο λόγο. Έχουμε τον οικονομικό κανονισμό και τους κανονισμούς που διέπουν τα ταμεία και τα γεωργικά ταμεία συμπεριλαμβάνονται εκεί. Μπορείτε έτσι επιγραμματικά να μας πείτε δύο-τρία στοιχεία κλειδιά για το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση της ανάπτυξης της υπαίθρου μέχρι την επόμενη ανανέωση της θητείας των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν μιλούμε τόσο για τις ενισχύσεις, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου ε, πραγματικά θα συνεχιστεί. Γιατί ξέρετε, η ανάπτυξη της υπαίθρου έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σαν το σιρτάρι στο οποίο βάζουμε όλα τα ξεχασμένα πράγματα ή όλα τα πράγματα τα οποία δεν έχουμε τι να τα κάνουμε και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να γίνει μια ε, σωστή ανάπτυξη της υπαίθρου από σήμερα μέχρι την επόμενη ημερομηνία αναθεώρησης της κοινή αγροτικής πολιτικής, της κοινή γεωργικής πολιτικής. Απάντηση. Σας ευχαριστώ κυρία Σέντερ, κυρία Γιάλα Σέντερ για τα ερωτήματα που μου θέσατε. Για τα ηθικά ζητήματα νομίζω ότι δύο ε, είναι αυτά που σας ενδιαφέρουν. Καταρχάς οι στατιστικές, άρα σε αυτό φαντάζομαι ότι θέλετε να σας δώσω αριθμούς υποθέσεων, δηλαδή πόσες υποθέσεις απασχόλησαν την Επιτροπή Ιδεοντολογίας και είδα ότι ε, θέσατε και ένα γενικότερο ερώτημα για την ιδεοντολογία. Για τα στατιστικά λοιπόν. Να σας πω ότι είμαι μέλος αυτή την Επιτροπή από τον Ιούλιο. Δηλαδή τρία, τρεις μήνες περίπου. Τον Ιούλιο εξελέγει και ανέλαβα αυτά τα καθήκοντα. Από τότε που έφτασα στην Επιτροπή Διοντολογίας, δεν είμαι βέβαιος, αλλά είχαμε 7 περιπτώσεις περίπου από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα. Περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου. Περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ καθηκόντων εντός ελεγκτικού συνεδρίου αυτή τη χρονική περίοδο και άλλων καθηκόντων που τα μέλη επιθυμούν να αναλάβουν. Επίσης, ε, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων πρώην μελών του ελεγκτικού συνεδρίου που θέλουν να ξεκινήσουν ξανά επαγγελματικές δραστηριότητες και ζητούν την άδεια του δικαστηρίου. Αυτές είναι οι βασικές ε, περιπτώσεις. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι Όταν βλέπουμε αυτές τις συγκρούσεις συμφερόντων και όταν θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει ζημιά στη φήμη και στο κύρος του ελεκτικού συνεδρίου, Μας ενδιαφέρει να κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ της του πραγματικού πλήγματος στο κύρος και του ε, ε, φαινομενικού πλήγματος στο κύρος, μεταξύ του ε, τωρινού και υπαρκτού ή υποθετικού. Ε, πράγματι πλήττεται το κύρος. Υπάρχουν διάφορες υποκατηγορίες δηλαδή και προσπαθούμε να κάθε περίπτωση να την κατατάξουμε αναλόγως. Αυτά για το πρώτο σας ερώτημα. Τώρα για την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ή την αναθεώρησή της θα έλεγα ότι εμείς είμαστε ελεγκτικός οργανισμός, ελεγκτική υπηρεσία και ο ρόλος μας είναι να κάνουμε δηλώσεις για τα ευρήματά μας, για τα γεγονότα. Επίσης ευθύνη μας είναι να ζητήσουμε από τον νομοθέτη να προσέξει ορισμένες πτυχές της υφιστάμενης πολιτικής και να την αναθεωρήσει και να τη μεταρρυθμίσει. Και σε αυτή την ε, ε, γραμμή θα κινηθώ. Εγώ είμαι ελεγκτής, βλέπω τα στοιχεία και τα γεγονότα μπροστά μου και μπορώ να δώσω ορισμένες ιδέες και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε την επόμενη χρονιά γιατί στο πρόγραμμα των εργασιών για την επόμενη χρονιά θα, κάνουμε, θα έχουμε ένα έγγραφο ενημερωτικό για τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Έχει έρθει η στιγμή να αξιολογήσουμε μία μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική και το σημαντικό είναι να έχουμε κριτήρια αξιολόγησης. Και όχι τόσο συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, η νέα πολιτική με βάση, βασίζεται στην αξιολόγηση. Η νέα πολιτική βασίζεται στα στοιχεία. Η νέα πολιτική έχει σταθερή και ισχυρή οικονομική βάση. Είναι δίκαιη. Ε, θυμάμαι την ερώτηση που μου έθεσε ο εισηγητής πριν. Η νέα αναθεώρηση της νέας πολιτικής είναι διαφανής, είναι απλή, είναι περιεκτική, με συνέπεια, με ολοκληρωμένη και υποπαρακολούθηση, εποπτευόμενη. Έχει αξιολογηθεί ο κίνδυνος που ε, συνεπάγεται. Αυτά είναι κριτήρια και είναι σημαντικά. Μπορώ να πω και περισσότερα πράγματα. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι στην αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πολιτική αυτή πρέπει για παράδειγμα να είναι στραμμένη προς την αγορά γιατί έχουμε ξεχωριστές δεσμεύσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Οκ. Okay. Άρα πρέπει να είναι μια πολιτική προσανατολισμένη προς την αγορά. Δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι σε αυτή την πολιτική πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες. Αλλά κάποια πράγματα να τα προσέξει περισσότερο ο νομοθέτης στο μέλλον. Π.χ η σχέση που ανέφερα προηγουμένως μεταξύ της γεωργίας και του περιβάλλοντος, διότι τα πράγματα δεν ε, λειτουργούν πολύ καλά. Και όπως είπε η κυρία Κρέσλε, έχουμε ε, εκθέση και θα τη στείλουμε στο Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι κάποιες ε, ιδέες Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητή της Επιτροπή θέλει να σχολιάσει γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι, θα ήθελα να πω το εξή. Τα τελευταία σας λόγια ε, μου, με κάνουν να σκεφτώ ότι βεβαίως πρέπει να υποστηρίξουμε τη βιώσιμη γεωργία αλλά και αυτές τις μικρές εκμεταλλεύσεις οι οποίες ε, σιγά σιγά ε, ε, χάνονται γιατί γνωρίζομαι και ότι οι αρρώσιμες γεές αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης πολύ συχνά και τις εποφαλμιούν διάφοροι των δικαιούχων ε, λαμβάνουν λιγότερο από 4.000 ε, ευρώ ε, και την ίδια στιγμή που οι μεγάλες εταιρείες παίρνουν εκατομμύρια. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Απάντηση. Αυτό είναι θεμελιώδες, βασικότατο ερώτημα για το μέλλον της ΚΑΠ. Σχετίζεται και με το ερώτημα του εισηγητού, τα δεοντολογικά, ηθικά ζητήματα. Τα στοιχεία, τα αριθμητικά που δώσατε μιλούν από μόνα τους. Αυτά είναι τα στοιχεία, το ξέρω, δεν τα αμφισβητώ. Και πιστεύω ότι κάποιοι μηχανισμοί θα πρέπει να υπάρξουν ε, στην ε, κοινή γεωργική πολιτική έτσι ώστε να αναθεωρήσουν και να διορθώσουν εν τέλει την κατάσταση γιατί διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα στο μέλλον και οι μικροί γεωργοί ε, ήδη, ήδη βρίσκονται σε κίνδυνο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ανταλλαγή απόψεων μαζί σας, αγαπητέ κύριε. Ε, σας ε, ευχόμαστε καλή τύχη και θα περάσουμε τώρα στην τελευταία ακρόαση. Είναι η ακρόαση της κυρίας Ιβάνοβα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην τελευταία ακρόαση. Καλωσορίσετε καλωσορίσατε αγαπητή κυρία και σας δίνω αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι ενώπιον σας ως ε, ε, υποψηφία από την Βουλγαρία για, το, για μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Επιτρέψτε μου να μιλήσω στη... Да благодаря на българското правителство за номинацията и доверието, които... Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση της Βουλγαρίας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και θεωρώ ότι είναι ένα μήνυμα που θέλει να δείξει ότι πραγματικά ε, θέλει, ότι χρειαζόμαστε περισσότερη δέσμευση στις θέσεις αυτές. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία του αιτήματο παράτασης ε, στη θέση μου ε, να σας πω τα εξής, να σας πω δύο λόγια για τις υψηλέγγους που έχω κάνει και τον τρόπο με τον οποίο θεωρώ ότι μπορούμε να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά τα αποτελέσματα και βεβαίως θα σας πω και ποιος, ποιοι είναι οι προσωπικοί μου στόχοι για μια ενδεχόμενη νέα ε, θητεία. Ε, έχω κάνει τέσσερι, ε, έξι, συγγνώμη, οκτώ ελέγχους, των οποίων ο κατάλογος πλήρως έχει υποβληθεί στην Επιτροπή. Έχουμε κάνει επίσης και τρεις εκθέσεις όσον αφορά την νεολαία και την απασχόληση, καθώς επίσης και την, το μηχανισμό Youth Guarantee και με τον τρόπο αυτό οδηγήσαμε τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να αναλάβουν περαιτέρω δράση έτσι ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των σημαντικών εργαλείων. Επίσης ε, ήμουν υπεύθυνη για το κεφάλαιο 6 ε, για 5 ε, συνεχή έτη και επομένως το κεφάλαιο 6 της ετήσιας έκθεσης ε, και με τον τρόπο αυτό λοιπόν ε, μπόρεσα να παίξω σημαντικό ρόλο ε, στο κατα... στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται το ελληνικό συνέδριο στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Βεβαίω, ε, η ετήσια έκθεση είναι το 50% της εργασίας. Ε, το επόμενο, το υπόλοιπο 50% είναι να βρούμε τον σωστό τρόπο να επικοινωνήσουμε τα ευρήματα σε όλους τους εμπλεκομένους. Από τη στιγμή που έφτασα στο ελληνικό συνέδριο ακριβώς προσπάθησα να μεγιστοποιήσω τον αντίκτυπο της εργασίας μας. Ξεκίνησα ας πούμε με την οργάνωση διαφόρων σημαντικών εκδηλώσεων ε, ας πούμε μια ε, διάσκεψη ε, ε, που κάναμε στις Βρυξέλλες με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Επίσης μια διάσκεψη πέρσι στο Λουξεμβούργο, περίπου 200 ήταν εκεί οι συμμετέχοντες ε, όσον αφορά την συνεργασία ε, με τα εθνικά συνέδρια και με τα άλλα όργανα. Εξαίρετη συνεργασία είχαμε με το Βουλγαρικό Ελεγκτικό Συνέδριο και όσον αφορά μεμονωμένους ελέγχους και όσον αφορά την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων οργανώσεων στη Σόφια για σειρά σημαντικών ε, θεμάτων και είμαι βεβαία ότι θα υπάρξουν ε, πολλές επιπλέον εκδηλώσεις και λόγω της επερχόμενης Βουλγαρικής Προεδρίας. Τα πιο σημαντικά στοιχεία πάντως τα οποία έχω να πω είναι, ε, αφορούν την σχέση με την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών. Εγώ έκανα πάντα, κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε πάντα να ε, ακολουθώ τις και να ακούω προσεκτικά τα σχόλιά σας γιατί αποτελούν πολύτιμες ιδέες για την μελλοντική μας εργασία. Καθώς επίσης να πω ότι είχα την χαρά να είμαι παρούσα στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, σε διερευνητικές αποστολές και αυτό είναι ένας πολύ καλός τρόπος ε, για να μπορέσουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα σε πέντε λεπτά να συνοψίσει κανείς την εργασία πέντε ετών. Ε, και θα ήθελα λοιπόν να σας πω τελειώνοντας ε, δύο λόγια για το πώς φαντάζομαι την μελλοντική θητεία. Βεβαίως απολύτως δεσμευμένη είμαι στις ε, βασικές αξίες ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Εάν η απόφασή σας για την παράταση της θητείας μου είναι θετική θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη θητεία αυτή έτσι ώστε να οικοδομήσω περαιτέρω επί των βάσεων που έθεσα τα προηγούμενα χρόνια. Θα συνεχίσω να προσπαθώ να διερευνώ ε, θέματα τα οποία είναι επίκαιρα και σημαντικά για όλους μας, ε, να βελτιώσω ε, εν τέλει την ποιότητα του παρεχομένου από εμά προϊόντος. Να σας πω επίσης ότι τα θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν τώρα είναι το η ευρυζωνικότητα ε, καθώς επίσης και η πρόσβαση μη αστικών περιοχών ε, σε νέες ε, τεχνολογίες. Οπουδήποτε διαπιστώνουμε ελλείψεις, οπωσδήποτε θα τις ε, αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε να δίνουμε ε, βέλτιστα παραδείγματα στην ε, διαχείριση των οικονομικών πόρων και με όλα αυτά σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει η Προεδρεύουσα, για την παρουσίασή σας. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Είχα το προνόμιο να παρακολουθήσω τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας μας στη Βουδαπέστη. Και αυτό ήταν πραγματική απόδειξη ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Η Επιτροπή μας με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ανέκαθεν ε, με συναρπάζει μια χώρα που ονομάζεται Βουλγαρία και το γεγονός ότι μια χώρα που ονομάζεται Βουλγαρία στέλνει γυναίκες και για το αξίωμα του Επιτρόπου και για το αξίωμα του μέλους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και θέλω να κάνω μια πρόβλεψη για σας. Ε, στην περίπτωση της Εσθονίας, το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου ε, ε, είχε, μπορεί και να έχει λαμπρή πορεία στην, και να ανέλθει μέχρι τον πρωθυπουργικό θόκο της χώρας. Ελπίζω να συμβεί και στη δική σας περίπτωση. Θα μου δώσει αυτό μεγάλη χαρά. Όμως, για να φτάσετε μέχρι εκεί πρέπει να απαντήσετε στο κάπως ε, ε, περίεργο ε, ερώτημά μου. Έχετε, φαντάζομαι ότι στο Λουξεμβούργο ίσως έχετε διαμέρισμα, αλλά εν πάση έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε έλεγχο στο Λουξεμβούργο στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αξιολογώντας αυτό το τωρινό σύστημα το οποίο επιβάλλει κάθε κράτος μέλος να έχει μια υπηρεσία, μια υπηρεσία να εδρεύει σε κάθε κράτος μέλος και κάθε κράτος μέλος να έχει έναν εκπρόσωπο, ένα, μια επίσημη θέση σε κάθε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι το ελεγκτικό συνέδριο ε, το πιο ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει μια ε, εύλογη και λογική μεταρρύθμιση της συμπεριφοράς και της δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για το ερώτημά σας. Έχουμε μια πολύ ανοιχτή και διαφανή διαδικασία στο πρόγραμμα εργασιών, πώς θα διαλέξουμε τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Είναι μια διαδικασία σε πολλά βήματα. Ε, τι κάνουμε κάθε φορά, κάθε χρόνο προσπαθούμε να ακούσουμε προσεκτικά, εγώ προσωπικά το πράτο, ε, τα σχόλια και τις προτάσεις σας και μετά τα συζητούμε με τους συναδέλφους εντός ελεγκτικού συνεδρίου και αποφασίζουμε συλλογικά ε, ποιο θέμα θα συμπεριλάβουμε στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Βεβαίως κάνουμε έλεγχο των θεσμικών οργάνων, των υπηρεσιών κάθε χρόνο. Αυτό εντάσσεται στο πεδίο ερμοδιοτήτων των συναδέλφων από το τμήμα 4 και θα τους το μεταφέρω. Σας διαβεβαιώ και θα το συζητήσουμε όταν συζητήσουμε το επόμενο μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών θα τους ενημερώσω ότι, ε, για το συγκεκριμένο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο συνάλφος κ. Σταϊκόφσκι παρακαλώ. Αγαπητή κυρία μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. τα γραφεία του ελεγκτικού συνεδρίου ε, σας αντιμετωπίζουν ως αστέρι. Ε, έχετε δυναμισμό ε, θετική ενέργεια. Και τώρα μοιάζεται σαν να σας ε, τυραννάμε. Μην μας φοβάτε, φοβάστε. Θα πρέπει να μας δείξετε την ενεργητικότητά σας ακόμα και αν έχουμε ε, δύσκολες, δυσάρεστες ερωτήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας ρωτήσω. Ε, είσαστε μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου εδώ και πέντε χρόνια. Ο προκάτοχός σας εδώ στην ακρόαση που διοργανώνουμε. Όταν το ρωτήσαμε για τις αδυναμίες ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, μας είπε ότι επειδή είναι μόνο ένα χρόνο στο ελεγκτικό συνέδριο, δεν έχει μπορέσει ακόμα να εντοπίσει αδυναμίες. Εσείς όμως είστε ήδη πέντε χρόνια στο ελεγκτικό συνέδριο. Έχετε δει λοιπόν κάποιες αδυναμίες. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι αδυναμίες αυτές και πώς ε, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτές τις αδυναμίες. Ε, πώς μπορείτε να βελτιώσετε την κατάσταση όπου ε, ίσως σε ποιους τομείς ε, θα θέλατε να εντοπίσετε και μη φοβάστε, δείξτε λιγάκι από τον ενθουσιασμό που σας χαρακτηρίζει. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που είπατε, αισθάνομαι λίγο αναστατωμένη γιατί είναι σαν να περνώ εξετάσει, αλλά δεν είναι και κακό αυτό, γιατί ειλικρινά λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου όλα σας τα σχόλια και ακούω πολύ προσεκτικά αυτά που μου λέτε, γιατί αυτή είναι και η πεμπτουσία της συνεργασίας μας. Αν δεν ακούει κανείς και νομίζω ότι τα ξέρει όλα, αυτό είναι πολύ κακό. Εγώ προσπαθώ να ακούω. Όσον αφορά τις αδυναμίες του συνεδρίου, Θέλω να σας πω, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πάντα μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Άσχετα αν είμαι 5, 6 ή 7 χρόνια στο ελεκτικό συνέδριο ή κάποιος άλλος, πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Και επιπλέον συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε σχετικά με τη στρατηγική μας για το 2020, 18 έως 2020 είναι προφανές ότι μπορούμε να εξορτολογήσουμε περαιτέρω τις εσωτερικές διαδικασίες του συνεδρίου, να βελτιώσουμε τις ετήσιες εκθέσεις, να αποδίδουμε περισσότερη, μεγαλύτερη σημασία σε θέματα απόδοσης. Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα που θέλω να εκπέμψω. Και βεβαίως ε, θα ε, εμφανιστώ και άλλες φορές στην Επιτροπή σας ε, μέχρι το τέλος του έτους και έχω την εντύπωση ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής ε, θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, δηλαδή πώς πρέπει να καταρτίζουμε τις αιτήσει εκθέσεις, γιατί τώρα προετοιμάζουμε τις αιτήσει εκθέσεις των επόμενων ετών και θα είναι λιγάκι διαφορετικές αυτές, γιατί θα λάβουμε υπόψη μας ένα νέο πλαίσιο, αλλά αλλαγές που έχουν επέλθει. Ε, θεωρώ ότι όπως σας είπα πάντα μπορεί κανείς να βελτιώνεται. Τουλάχιστον αυτό εγώ έτσι το αντιμετωπίζω. Ο συνάδελφος ε, Άλλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για τον διορισμό σας και θέλω να σας πω ότι εμείς χαίρομαι που συμβάλλουμε ε, στο ότι συμβάλλουμε στην ε, ισότητα των δύο φίλων στο ελεγκτικό συνέδριο. Ε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και όπως είπατε είσαστε για πέντε χρόνια στο ελεγκτικό συνέδριο και ασχολείστε με την οικονομική, κοινωνική, εδαφική συνοχή και θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Από την αρχή της ε, περίοδου του προγράμματος νομίζουμε ότι θα έπρεπε να ληφθούν περισσότερα μέτρα στα κράτη-μέλη για την κοινωνική συνοχή. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις θα εξισορροπηθούν αυτές στο πλαίσιο του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και κατά την άποψή σας πώς θα επηρέαζε αυτό τα ποσοστά ασφάλματος Και έχω και άλλη μια ερώτηση που αφορά στην απασχόληση των νέων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέσα του 16 η ανεργία των νέων ήταν περίπου 18,8%. Και αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια εκ μέρους των νέων. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για την ποιότητα των προγραμμάτων που επιλέγονται για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας. Η πρώτη αφορά το ποσοστό σφάλματος και την απορρόφηση. Ποσοστό σφάλματος είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση ε, βλέπουμε ότι με την πάρδο των ετών μειώνεται κατά το ποσοστό σφάλματος. Ε, είχαμε, είχαμε διψήφια στοιχεία, 11 περίπου 100 και φτάσαμε στο 4,8% το 16%. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σας πω ότι είναι πάνω από το όριο του 2%. Ε, και αυτό έχει κυρίως σχέση με ότι υπάρχουν προβλήματα στη γεωργία τα αίτια των σφαλμάτων, όπως σας είπα, περίπου το ίδιο γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή, μη επιλέξιμες ε, δαπάνες, ε, μη επιλέξιμη δικαιούχη παραβίαση εθνικών κανόνων στα κρατικά επιδόματα και στους δημόσιους διαγωνισμούς, στις κρατικές προμήθειες. Αυτά, ε, είναι, αυτά επηρεάζουν περισσότερο από όλα τα ποσοστά ασφάλματος. Τώρα, όσον αφορά την χαμηλή απορροφησιμότητα, εμείς ε, ως ελεγκτές θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν θέλω όμως να προκαταλάβω τίποτα για το ποιο θα είναι το ποσοστό σφάλματος κατά τα επόμενα έτη. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Όμως το θέμα της απορρόφησης ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, το έχουμε ήδη πει και πέρυσι αλλά και φέτος στην ετήσια έκθεση ότι η απορρόφηση είναι πολύ χαμηλή μόνο το 77% ε, έχει απορροφηθεί το 16% και αυτό αυτό ε, προφανώς ε, θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην εφαρμογή. Και δράδω με τις ευκαιρίες για να σας πω ότι ε, θέλουμε να υπάρχει μια ειδική έκθεση για την απορρόφηση. την, έχει αναλάβει ένας άλλος συνάδελφος στο δεύτερο τμήμα, σε άλλο τμήμα. Νομίζω στις αρχές του επόμενου αετούς θα δημοσιευτεί η έκθεση αυτή και εκεί θα υπάρχει λεπτομερέστερος σχολιασμός για το θέμα της απορρόφησης. Για την ανεργία των νέων. Προφανώς αυτό είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ε, τρεις εκθέσεις έχουμε για αυτό το θέμα. Ξεκινήσαμε με τον έγκαιρο σχεδιασμό, ε, να δούμε λιγάκι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τι ακριβώς κάνει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σχεδιασμό των ε, προγραμμάτων και εκεί εντοπίσαμε τρεις βασικούς κινδύνους στην εφαρμογή. Πρώτον, ανεπάρκεια κονδυλίων. 12,5 δις διατίθενται για την αγγίηση των νέων και για τη σχετική πρωτοβουλία. Και με βάση ανεξάρτητους οργανισμούς και ελέγχους γνωρίζουμε ότι θα πρέπει κάθε χρόνο να ε, δαπανώνται περίπου 45 με 50 δισεκατομμύρια κατέτος για την ανεργία των νέων. Άρα υπάρχει έλλειψη εδώ. Και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι μετά ε, κάναμε μία δεύτερη έκθεση για την ε, εγγύηση για τους νέους. Τα αποτελέσματα στα κράτη-μέλη τα ελέγξαμε. Πράγματι διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος ότι υπήρξε ε, πρόοδο στα επτα κράτη-μέλη που επισκεφτήκαμε, αλλά ακόμα υπολείπονται αρκετά και πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι που τόσο στην Επιτροπή ε, και στις δύο εκθέσεις, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ε, τεκμηριωμένες προσδοκίες για να μην απογοητευτούν οι νέοι στο μέλλον. Γιατί αν συμβεί αυτό δεν είναι καλό ούτε για τους ίδιους, ούτε για μας, ούτε για την Ευρώπη. Άλλοι έξι συνάδελφοι θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις, που σημαίνει ότι στις ερωτήσεις ε, θα πρέπει ε, να περιστούμε στο ένα λεπτό, στις απαντήσεις δύο λεπτά και θα τα καταφέρουμε να τελειώσουμε με αυτό το σύστημα στις 11.30. Ευχαριστώ. Ε, Δουλεύουμε πολύ στενά για το θέμα του Youth Guarantee και Youth Initiative. Και γι' αυτό δεν θα ρωτήσω για αυτά. Κάτι γενικότερο θα ρωτήσω. Οι συνάδελφοι ανέφεραν την ε, καθοδική τάση των συχνοτήτων λάθους, ε, συχνοτήτων σφαλμάτων, error rates. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί πιστεύετε ότι είναι πιο θετική η στάση αυτή. Ε, έχει αλλάξει η στάση των ελεκτών. Με ποιο τρόπο. Εν συντομία, ναι πράγματι είναι καθοδική η τάση, όμως θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Είμαστε πάνω από το 2%, άρα δεν είμαστε ιδανικό. Ε, το 4,8% είναι λίγο και λιγότερο από το παρελθόν, αλλά συνεχίζει να είναι πάνω από το 2%. Τους λόγους νομίζω τους ανέφερε ο πρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου. Υπάρχουν και στην ετήσια έκθεση Φέτος έχουμε τις μισές πληρωμές από αυτές που δικαιούνται οι αγρότες και άρα όλα αυτά, ε, οι μισές είναι κάτω από το materiality threshold, κάτω από το 2%, οι άλλες μισές είναι πάνω από το 2% και στο, στα θέματα συνοχής ε, διαπιστώνουμε μείωση των error rate και στις δημόσιες αγορές και σε διάφορους ε, κρατικές ενισχύσεις, στους διαγωνισμούς. Όλα αυτά σχετίζονται και με τις συστάσεις μας. Έχουμε βελτιώσεις και στις, στους ελέγχους που κάνουν οι αρχές των κρατών μελών αλλά και στους ελέγχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί αθρηστικά εξηγούν γιατί για πρώτη ε, φορά ε, φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Η κυρία Γιαμπάγιοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία ε, η, Ιβάνοβα, ε, μην ε, ε, ασχολείστε με το συνάδελφο, σας ζηλεύει γιατί έχουμε τόσους πολλά μέλη από τη Βουλγαρία παρόντα, ενώ εμείς είμαστε οι μόνοι δύο Τσέχοι που προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, Σα συγχαίρω. Θεωρώ ότι το θέμα της εγγύησης για τους νέους είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Η ανακοίνωση επίσης ε, που ενισχύει τον αντίκτυπο της δουλειάς του ελεκτικού ε, συνεδρίου στους Ευρωπαίους πολίτες είναι κάτι το πολύ καλό και σας ευχαριστώ και γι' αυτό. Μας ενδιαφέρει ε, το γεγονός ότι δίδεται έμφαση πλέον στην απόδοση, στις επιδόσεις και υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες και συγκεκριμένα αποτελέσματα αλλά οι δείκτες και τα αποτελέσματα δεν ασχολούνται με την βιωσιμότητα του συστήματος και τη μελλοντική αποτελεσματικότητα. Δηλαδή είναι πράγματα που έχουν προστιθέμενη αξία αλλά δεν μπορούν να φανούν αμέσως. Άρα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία στους δείκτες που έχουν να κάνουν με τις επιδόσεις και για τα άμεσα τα αποτελέσματα και μεταξύ αυτών και μεταξύ των μελλοντικών και της προστιθέμενης αξίας που θα δημιουργηθεί απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Για το θέμα της επλούστευσης πρέπει να συζητήσουμε ποιο ρόλο θα έχουν οι δείκτες αποδόσεων και επιδόσεων και αποτελεσμάτων. Είναι πολύ της μόδας ο όρος, αλλά να μην και το, το παρακάνουμε κιόλας. Θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση. Έχουμε μια πολύ καλή δική έκθεση που έχει ήδη δημοσιευθεί, είναι διαθέσιμη την έκθεση για τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης Ο ρόλος λοιπόν των δικτών για τα αποτελέσματα και ο τρόπος με τον οποίο έχουν μπει, ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη-μέλη προσπαθούν να καλλιεργήσουν την κουλτούρα των αποδόσεων και επιδόσεων θεσπίζοντας τόσους πολλούς δείκτες μας έχουν οδηγήσει να έχουμε χιλιάδες δείκτες σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο περιφέρειας άρα φτάνουμε σε ένα σημείο που τελικά μπερδευόμαστε τι είναι αυτό που μετράμε πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτή την πληροφόρηση αθρηστικά και ποιο νόημα βγάζει. Και αν εναρμονιστούν αυτές οι, αυτοί οι δείκτες, ε, σε ποιο αποτέλεσμα θα οδηγηθούμε. Άρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, να είμαστε προσεκτικοί ποιου δείκτες θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε, ποιου δείκτες θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε γιατί δεν χρειάζονται, ποιε είναι οι καλές πρακτικές που θα πρέπει να διαδίδονται και η Επιτροπή, ξέρετε, παρουσιάζει τις νομοθετικές προτάσεις σε σωστές χρονικές στιγμές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην έχουμε επιπλοκές στο μέλλον. Με δύο λόγια λοιπόν να σας πω ναι στους δείκτες αλλά όχι με κάθε τίμημα να τους χρησιμοποιούμε αλλά τους σωστούς, τους καλούς δείκτες που θα μετρούν τα σωστά πράγματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Ιβανόβα για την παρουσίασή σας. Με μεγάλη προσοχή έχουμε ε, διαβάσει την τροχιά που ακολουθήσατε ε, και βεβαίως και τις ε, πολλές εκθέσεις τις οποίες έχετε συντάξει. Μία συγκεκριμένη ερώτηση για το μέλλον ήθελα εγώ. Βρισκόμαστε εν μέσω προβληματισμού για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά αυτό αγγίζει και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων και το ελεγκτικό συνέδριο. Πώς θα βλέπατε εσείς ε, το ελεγκτικό συνέδριο τα επόμενα έξι χρόνια επί τη βάση της εμπειρίας την οποία έχετε ε, πλέον λόγω της ε, προηγούμενης ε, θητείας σας. Θα θέλαμε και σε χοντρές αδρές γραμμές να μας κάνετε μια παρουσίαση γιατί σε, πέντε λεπτά, σε δύο λεπτά συγγνώμη, δεν είναι δυνατόν να μας τα πείτε όλα. Απλώς ποιος είναι ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου που δεν, είναι, δεν αφορά πλέον μονάχα τα MFF αλλά ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Σαλαφράγκα. Ε, το ανέφερα αυτό ε, στην αρχική μου παρουσίαση αλλά ξεπερνούσε μετά τα πέντε λεπτά και το έκοψα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα φυσικά και θα ήθελα και εγώ να σας πληροφορήσω για τις προσωπικές μου απόψεις όσον αφορά τις τάσεις και τις κατευθύνσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Βεβαίω υπάρχουν στοιχεία αντικειμενικά, ζητήματα προτεραιότητα, ε, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Στεχόφσκι στην ερώτησή του. Βρίσκονται αυτά όμω και στην ιστοσελίδα του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, αλλά αν θέλετε να τα επαναλάβω, ναι, νομίζω ότι είναι ε, σημαντικό να ευθυγραμμίσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες έτσι ώστε να επικεντρωθούμε σε θέματα, στο θέμα της αποδοτικότητας και της απόδοσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερες εκθέσεις αποδοτικότητας αλλά καλύτερη ε, αναφορά καλύτερης ποιότητας επομένως ε, εκθέσεις ε, αποτελεσματικότητας. Αυτές θα έχουν καλό αντίκτυπο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο σχόλια ένα σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρατε όσον αφορά την συνοχή της ετήσιας έκθεσης. Ε, δεν ξέρω πόσο μπορείτε να μας απαντήσετε βέβαια, αλλά ποια ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος η αιτία της χαμηλής απορροφητικότητας των διαρθρωτικών πόρων. Επίσης, όσον αφορά την ψηφιοποίηση και το ψηφιακό θεματολόγιο, δεν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια σύγκρουση συμφερόντων γιατί στην Κομισιόν Έχετε την κυρία Γκάμπριελ ως ε, ε, συνομιλητή που είναι από τη χώρα σας και από το κόμμα σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα. Σας ακούω εσάς ειδικά πολύ προσεκτικά και με μεγάλη προσοχή λαμβάνω υπόψη μου τα σχόλιά σας. Όσον αφορά το θέμα της συνοχής, ε, η αποτελεσματικότητα του naming and shaming Κοιτάξτε, από όταν ήμουν μέλος της Επιτροπής ε, το θέμα ήταν επίκαιρο. Εγώ θα το θα το έθετα διαφορετικά. Πρέπει να έχουμε περισσότερη γεωγραφική ας πούμε, θεώρηση. Όσο, όσο περισσότερες αντικειμενικές πληροφορίες ε, και όσο πιο διάφανες είναι οι πληροφορίες ή ο τρόπος ε, αναφοράς τους είναι το, τόσο το καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε ίσως στη συζήτηση για την επόμενη απαλλαγή. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι, αλλά ενδεχομένως να είμαστε σε θέση να δώσουμε πιο πολλές ε, πληροφορίες ε, ε, που θα βασίζονται σε γεωγραφικές εκτιμήσεις. Αλλά έχουν γίνει αλλαγές γενικά και στους ε, συστήματα ελέγχων της ε, Κομισιόν ε, φέτος, γιατί από αυτήν την χρονιά και μετά θα έχουμε ετήσιο κλείσιμο των λογαριασμών και η Κομισιόν δέχεται, θα δέχεται ε, πλέον τους λογαριασμούς μονάχα εάν ε, το ποσοστό λάθος είναι κάτω από το 2% και ε, θα υπάρχει και ένα υπόλοιπο που θα διακρατείται της τάξης του 10% σε αντίθετη περίπτωση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία αυτά, ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τον τρόπο εργασίας μας. Και αν αυτό λειτουργήσει θετικά, θα είμαστε σε θέση, νομίζω, και ενδεχομένως αυτό θα αποτελέσει άλλωστε και ένα από τα κεντρικά στοιχεία της πιλωτικής προσέγγισης. Τότε, λέω, θα είμαστε ενδεχομένως σε θέση να δώσουμε ε, πληροφορίες ε, σε σχέση με γεωγραφική κατανομή. Ε, Βεβαίω δεν μπορούμε να καλύψουμε τα 28 κράτη. Θα επιλέξουμε 5-6 κράτη-μέλη σε κάθε ειδική ε, έκθεση για την Youth Guarantee. Νομίζω ότι ε, ε, είχαμε 7 μάλιστα, είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των κρατών. Όσον αφορά το ψηφιακό θεματολόγιο, δεν είχα καν σκεφτεί το ενδεχόμενο σύγκρουση συμφερόντων γιατί το θέμα αυτό άρχισε να με απασχολεί πολύ παλιότερα και σίγουρα πριν να είναι ε, η συγκεκριμένη επίτροπος ε, ε, στην συγκεκριμένη θέση. Ξεκινήσαμε πολύ καιρό πριν και τώρα προετοιμάζουμε το πρώτο προσχέδιο έκθεσης και δεν νομίζω ότι μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η εργασία των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου διακρίνεται πάντα από διαφάνεια ε, και το ελεγκτικό συνέδριο συλλογικά ε, αναθέτει ένα μέλος ε, μια συγκεκριμένη έκθεση και μένα μου ανατέθηκε η έκθεση αυτή έχει υπάρξει αυτή η σύμπτωση ε, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Δεν νομίζω πάντως ότι ε, θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά που υποβάλλατε το ερώτημα αυτό. Και εγώ έχω βάλει τον εαυτό μου στον κατάλογο των ομιλητών με την ερώτηση που κάνω, έκανα σε όλους ε, τους υποψήφιους, ε, ε, αν έχετε σπίτι στο Λουξεμβούργο, πόσο συχνά εργάζεστε ή είστε παρούσα στο ελεγκτικό συνέδριο και σχετικά με αυτό που είπε η κυρία Αγιάλα Σέντερ για τις εκθέσεις ε, αναχώρα. Εμείς δεν το σκεφτόμαστε οτι ότι είναι endo-shaming ή naming, αλλά ε, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πληροφορίες, έγγραφα που ε, υπάρχουν και πληροφορίες αυτά να χορηγούνται, να δίδονται στο ελεγκτικό συνέδριο, να ε, συντονίζονται, να ελέγχονται, να επανελέγχονται. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μας. το είδαμε ήδη να συμβαίνει αυτό και νομίζω ότι εκεί που συνέβη ε, μπορέσαμε να έχουμε καλύτερη εικόνα για τα προβλήματα της ε, χώρας, κυρίως ε, στο θέμα των κρατικών προμηθειών. Ίσως μπορείτε να τοποθετηθείτε, να μας πείτε αν τελικά το ελεγκτικό συνέδριο θα μας στηρίξει σε αυτό το έτοιμά μας για τις κρατικές προμήθειες και για τις αιτήσεις εκθέσεις. Όχι, εγώ δεν έχω διαμέρισμα στο Λουξεμβούργο. Ζω στη Γερμανία, στα σύνορα με το Λουξεμβούργο. Ε, πηγαίνω όμως κάθε μέρα στο Ελληνικό συνέδριο. Ο γιος μου πηγαίνει ε, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο που είναι κοντά στο ελεγκτικό συνέδριο. Άρα δηλαδή είμαι παρούσα, συνέχεια παρούσα ε, στο ελεγκτικό συνέδριο. Η δεύτερη μου ερώτηση για τις ε, εκθέσεις αναχώρα. Γνωρίζω πολύ καλά τοποθέτησή και τα έχω ήδη μεταφέρει ε, στην ε, συζήτηση. Τα έχω ήδη μεταφέρει στους αδέλφους. Ε, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα και εγώ τότε να πάμε μαζί αυτή την αποστολή γιατί και για μένα ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η επίσκεψη. Επισκεφτήκαμε από κοινού την Αγέν και μετέφερα ε, τα σχόλια στο συνάδελφό μου που ήταν αρμόδιος για την σύνταξη της έκθεσης. Και περιμέναμε ανυπομονησία και τη δική σας την έκθεση για αυτή την επίσκεψη, γιατί θα μας βοηθήσει να έχουμε και εμείς καλύτερες ιδέες. Τώρα, για την Ουγγαρία δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί αυτό θα πρέπει να είναι απόφαση του ε, συνεδρίου. Αλλά σας υπόσχομαι ότι θα σας ενημερώσω το των δυνατών, το τι αποφάσισε το δικαστήριο μάλλον ε, και βεβαίως είμαι και απολύτως στη διάθεσή σας ε, να συνεργαστούμε. Ε, τελευταίος, ο συνάδελφος Νόβακοφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάντα πίστευα ότι αν κάποιος ε, υποβάλει υποψηφιότητα για δεύτερη φορά, δεν χρειάζεται πολλά λόγια, γιατί μιλούν οι πράξεις του. Έτσι λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, ποια πρωτοβουλία σας κρίνετε την πιο αξιόλογη και την πιο σημαντική. Και δεύτερον, τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε για να προάγετε τις δραστηριότητες του συνεδρίου σε διάφορα κράτη-μέλη, γιατί ο ρόλος του συνεδρίου υποτιμάται σε πολλά κράτη-μέλη και οι πολίτες δεν γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνει το Ελληνικό Συνέδριο για να προστατεύσει τα ε, συμφέροντά τους. Uh, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι ανέφερα ήδη την εγγύηση για τους νέους. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα, ένα από τα πιο σημαντικά οικονομικά εργαλεία, πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Θεωρώ ότι ε, αυτό το πρόγραμμα έχει αληθινό αντίκτυπο στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Ε, όταν δημοσιεύσαμε το πρώτο έλεγχο, ε, σε σχέση με τον ορισμό δεν είχαμε πει πολλά, ούτε είχαμε κάνει πολλά, ούτε είχαμε ορίσει το τι είναι το good quality offer, μία προσφορά καλής ποιότητας. Και μετά από την έκθεσή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πιο λεπτομερείς ε, οδηγίες ε, για τα κράτη-μέλη, δεν σημαίνει ότι το ορίσαμε νομικά, αλλά δώσαμε περισσότερα κριτήρια, περισσότερους χαρακτηρισμούς ε, που θα μπορούσαν να πλαισιώσουν αυτή την έννοια της προσφοράς ε, καλής ποιότητας για να μην αναγκάζονται οι νέοι τελικά να έχουν μια προσφορά για λίγες μέρες, για δύο εβδομάδες και μετά ξανά πάλι ε, στο δρόμο να ψάχνουν. Τότε επίσης παρατηρήσαμε ότι δεν είχε προβλεφθεί λογοδεσία η αναφορά των λογαριασμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εμείς στην έκθεσή μας το είπαμε αυτό. Και στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε επιθύμως, επισήμως να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ε, αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις συζητήσεις και τις αποφάσεις στο πλαίσιο του ΕΜΚΟ. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός αντίκτυπος. Τώρα, για το ρόλο του δικαστηρίου στα κράτη-μέλη, νομίζω ότι έχουμε κάποια παραδείγματα, τα παρουσίασα με το κράτος μέλος που γνωρίζω περισσότερο και αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί βέβαια και στο μέλλον. Δεν περιορίζομαι στο κράτος μέλος που γνωρίζω περισσότερο από όλα, αλλά και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη όπου με προσκαλούν προσπαθώ να προωθώ το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου με τον Λιθουανό συνάδελφο έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία και ε, προωθούμε αυτή την εκδήλωση για την προώθηση της έκθεσης για τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά εργαλεία την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς ε, και έτσι φτάσαμε στο τέλος της ακρόασης. Ε, θα ήθελα λοιπόν όλοι όσοι δεν είναι μέλη ή σύμβουλοι να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο την ψηφορία. Επιτρέψτε μου να πω το εξή για άλλη μια φορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τα μέλη αλλά και όλους τους συμβούλους και συνεργάτες από τις πολιτικές ομάδες γιατί μας βοηθάνε να κάνουμε τη δουλειά μας και κυρίως απευθύνομαι στη γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ.